Uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω ότι αύριο στην πρωινή μας συνεδρίαση έχουμε στο πρόγραμμά μας την έκθεση του κυρίου Ταγιάννη για, την, ε, για το αποθεματικό σταθεροποίησης της αγοράς ETS Αύριο το πρωί η έκθεση του κυρίου Ταγιάννη. Πρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμα και την έκθεση του κυρίου Ταγιάννη για την ε, σταθερότητα της αγοράς και το αποθεματικό στην απογευματινή συνεδρία, δηλαδή το πρωί αύριο θα ολοκληρώσουμε περίπου στις 11.30, δηλαδή νωρίτερα. Και η απογευματινή μας συνεδρίαση θα έχει ως πρώτο σημείο το 13, η έκθεση του κυρίου Ντεμπάκερ, ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες, μετά, μετά τον κύριο Ντεμπάκερ, ο κύριος Ταγιάννη, αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς, για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αεριού θερμοκηπίου. Και έχουμε και τον δόκτορα Ρούσνακ, το σημείο 12. Η σειρά της απογευματινής συνεδρίασης, 13, Ντεμπάκερ, 11 έκθεση τα Γιάννη και 12 Διεθνής Χάρτης Ενέργειας 2015. Αυτά για την ε, αυριανή συνεδρίαση. Και να θυμίσω ότι σήμερα στις 6.30 μετά την συνεδρίαση θα έχουμε την χριστουγεννιάτικη δεξίωσή μας. Ελπίζω να μείνετε όλοι ως τις 6.30. Δηλαδή 3.30 ώρες. Ωραία. Πρώτο σημείο λοιπόν της απογευματινής μας συνεδρίασης. Σημείο 5. Έχουμε πολλά σημεία μπροστά μας. Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εξεχρονισμού του δημόσιου τομέα. Να σας θυμίσω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαλειτουργικότητα, για το δεύτερο πρόγραμμα, η δεύτερη πρόταση, θέλει να, ε, να δώσει συνέχεια στο πρόγραμμα που λύγει την, ε, στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Το Δημοσιονομικό Χαρτοφυλάκιο για την ε, προκοδότηση του δεύτερου προγράμματος 2016-2020 για πέντε χρόνια είναι 130 ε, εκατομμύρια ευρώ περίπου. Και τώρα θα συζητήσουμε, να θυμίσω σε όλους, Έχουμε εισηγητή, τον κύριο Κάρλους Ζουρίνιου, που είναι εδώ και θα σας παρακαλέσω, συνάδελφε, να ξεκινήσετε. Να ξεκινήσετε με την παρουσίασή σας. Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας για την πρόταση της Επιτροπής. Το δεύτερο πρόγραμμα για τη διαλειτουργικότητα. Κύριε Ζωρίνιου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως μόλις είπατε, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του προγράμματος ΙΖΑ, του προγράμματος ISA που θα ισχύσει στο τέλος του 2015. Το πρόγραμμα αυτό ανοίγει ένα νέο κύκλο και παρόλο που είναι ένα πρόγραμμα που απλώς συνεχίζει το προηγούμενο, πρέπει να λάβει υπόψη και τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν συμβεί μεταξύ. Πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις νέες ανάγκες των δημοσίων δικήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και τις νέες ευκαιρίες του cloud computing του υπολογιστικού νέφους. Θα ήθελα εδώ να τονίσω το ρόλο των επιχειρήσεων και των πολιτών που είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος αυτού. Το προηγούμενο πρόγραμμα επικεντρωνόταν στην ε, ε, αμοιβεοποίηση και στη συνεργασία των δημόσιων δικήσεων. Τώρα, ο εξυγχρονισμός των δημόσιων δικήσεων πρέπει να φτάσει και στους πολίτες. Αυτός είναι ο στόχος του δεύτερου προγράμματος. Τα που θα ορίσουμε εμείς ως κριτήρια για την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος και όχι μόνο από την πλευρά της προσφοράς αλλά και της ζήτησης θα είναι καθοριστικά. Δηλαδή, τη δυνατότητα των δημόσιων δικήσεων, του δημόσιου τομέα, να δώσει περισσότερες απαντήσεις και πιο αποτελεσματικές απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών. Η διαλειτουργικότητα, είναι πάντοτε στην καρδιά της λειτουργίας των δημοσίων διοικήσεων και θα έπρεπε να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των πολιτών. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια απόφαση όχι τόσο τεχνοκρατική, αλλά με την Ευρώπη που θέλουμε να περάσει σε ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της ψηφιακής μας ατζέντα, του ψηφιακού θεματολογίου για τη στήριξη των δημόσιων διοικήσεων στην Ευρώπη, και αυξάνει το δυναμικό ώστε οι δημόσιες δικήσεις της Ευρώπης να λειτουργήσουν ως φορείς θετικής ε, συνεισφοράς στην ποιότητα της οικονομικής μας παραγωγής και το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων, των πολιτών. Πιστεύω ότι η απόφαση αυτή είναι καλή στη βάση της, είναι σωστά διαφρομένη, σωστά τεκμηριωμένη, αλλά μπορεί ε, επιπλέον και αυτή θα είναι η δική μας συμβολή του Ευρωκοινοβουλίου να δώσει περισσότερη έμφαση στην οικονομική και κοινωνική ανάληψη ευθύνη για το πρόγραμμα. Ε, εδώ προτείνω 7 γραμμές για να το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την κοινή γλώσσα που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε εδώ. Θέλουμε η ευρωπαϊκή οικονομία να είναι πιο ανταγωνιστική. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα σύνολο, ένα καταπίστευμα για να το πω έτσι, ε, λύσεων και προτάσεων, τα, οι οποίες να μπορούν να αξιοποιηθούν στα νέα προγράμματα. Τα νέα προγράμματα χρήζουν νέας ερμηνείας, επειδή έχουν προκύψει εδώ μεταξύ νέες εξελίξεις και η πλατφόρμα Join Up καθώς και η νέα θηρίδα είναι στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιώσεις. Με την τεχνολογική επανάσταση και τις σημερινές προκλήσεις πρέπει να διαφυλάξουμε καλύτερα τον ιδιωτικό βίο και την ασφάλεια υπό την σκοπιά των επιχειρήσεων και των πολιτών. Επίσης, παρόλο που δεν είναι από τα βασικά προβλήματα του προγράμματος ΙΖΑ, επίσης μπορούμε να απλοποιήσουμε τις επενδύσεις και το πεδίο που θέλουμε να καλύψουμε με αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να, δείξουμε ενδιαφέρον για, για τα κίνητρα εντατικοποίηση της συνεργασίας. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σωστή κατανομή των ευθύνων του προγράμματος μεταξύ των 28 χωρών με 130 εκατομμύρια που ανέφερε ο πρόεδρο ε, η κάθε χώρα θα λάβει το δικό της ε, τμήμα από τα κονδύλια, όμως πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει και διαδικητική συνεργασία. Όσο, περισσότερο συνεργασία, όσο περισσότερη συνεργασία πετύχουμε, τόσο πιο ε, αποτελεσματικές θα είναι οι, θα είναι οι μορφές λειτουργία του προγράμματο. Επίση, πρέπει να ασχοληθούμε με την ικανοποίηση των ε, πελατών εντό εισαγωγικών, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Θα πρέπει αυτό το στοιχείο να χρησιμοποιηθεί για την συνολική αξιολόγηση του προγράμματο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρο. Ευχαριστώ, συνάδελφε και όντε εισηγητέ τώρα από το ΕΛΚΑ. Ο κύριο Μπόνι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πολωνικά. Το πρόγραμμα αυτό, το ΙΖΑ 2, θα μειώσει το διοικητικό κόστος. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγαράς θα βοηθήσει τη ροή προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς ε, διοικητικά και λοιπά εμπόδια και θα καταστεί πιο αποτελεσματικό το σύστημα, εφαρμόζοντας ε, μεγαλύτερο τμήμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ασφαλώς μπορεί να διαδραματίσει ρόλο κλειδί, βελτιώνοντα την ενιαία ψηφιακή αγορά που αποτελεί μια προτεραιότητα. Τα οικονομικά ωφέλη είναι σαφή. Οι σχέσεις ε, της κυβέρνησης των κρατικών υπηρεσιών με του ε, πολίτες ε, ή σε ό,τι αφορά τη διάσταση του εμπορίου μεταξύ των διάφορων τομέων το ΙΖΑ 2 καλύπτει διάφορους τομείς όπου χρειάζεται διαλειτουργικότητα και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ποιες είναι λοιπόν οι απειλές σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Καταρχάς έχουμε το θέμα του χρόνου. Αν το πρόγραμμα δεν είχε εγκριθεί, αν δεν, ήταν, αν δεν σκοπεύαμε να εγκρίνουμε τα μέτρα συντονισμού θα αυξάνονταν το κόστος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον πολίτη. Μία σειρά διαφορετικών λύσεων θα οδηγούσε σε όλο και πιο πολλά εμπόδια, τα οποία θα ήταν δύσκολο να ξεπεραστούν. Γι' αυτό ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή του προγράμματος θα ολοκληρωθεί το 2015 προκειμένου να ξεκινήσει το 16. Σημαντικό είναι επίσης να συγχρονιστούν οι δράσεις μεταξύ της, του Connecting Europe Facility και του ISA 2, γιατί μπορεί να υπάρχει κάλυψη μεταξύ των δύο προγραμμάτων. Η υπηρεσία μηχανικής μετάφρασης για τις χώρες των κρατών μελών, το πρόγραμμα αυτό, υποτίθεται ότι θα αντιτίθεται δωρεάν ως τμήμα του ISA 2, ενώ στο Connecting Europe Facility υπάρχει ένα σύστημα οικονομικής ε, εφαρμογής για τον ίδιο σκοπό. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει αυτή την αντίφαση που φαίνεται να υπάρχει. Ύστερα υπάρχει το θέμα της επιβεβαίωσης των έργων υπό το πλαίσιο του ΙΖΑ 2 για τα επόμενα χρόνια. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πώς πρόκειται να οργανώσει το ζήτημα αυτό η διαλειτουργικότητα καλύπτεται από το ΙΖΑ 2 που θα ορίσει και το μορφότυπο για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Τι περαιτέρω βήματα προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εφαρμόσει το σύστημα αυτό. Υπάρχει και το ψηφιακό ζήτημα. Και αναρωτιέμαι μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ε, προετοιμάσει ένα κανονισμό το οποίο θα βελτίωνε την κατάσταση. Θα έλυνε πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη συνοριακή και την ηλεκτρονική άσκηση δημοσίων υπηρεσιών για να ολοκληρωθεί και η ενιαία αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρότεινα λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε να προετοιμάσουμε το, συντομότερο δυνατό το σχέδιο αυτό για να επιλύσουμε και το πρόβλημα, τα προβλήματα που ανέφερα. Σας ευχαριστώ η κυρία Κάλλας η οποία αντικαθιστά τον κύριο Τόιρερ, σκιώδη εισηγητή τη Άλντε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να δείξω μερικά σημεία. Είναι σημαντικό το πρόγραμμα ΙΣΑ να λάβει υπόψη και τις προθεσμίες που έχουν οριστεί σε διάφορους τομείς σε ό,τι αφορά την εκτονικές Διαγωνισμού, για παράδειγμα, θα πρέπει να καταστεί αυτό ο κανόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο δεν ισχύει σήμερα. Προθεσμία για την εκτέλεση αυτή του προγράμματος είναι τα μέσα του 2015. Υπάρχει λοιπόν κατεπίγουσα ανάγκη διαλειτουργικότητας. Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά τελωνία, το e-customs, σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές υποθέσεις, τις θεωρήσεις, Schengen, η νέα η υπηρεσία που χειρίζεται τα συστήματα αυτά θα μπορούσε να υιοθετήσει το κοινό σύστημα πληροφορικής για τα τελωνία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δώσουμε στο ίσα ε, επιπρόσθετα κατοίκοντα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει εμπιστοσύνη στα ψηφιακά, στις ψηφιακές λύσεις. Και εδώ σημαντική είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και δεν εννοώ την ασφάλεια των δεδομένων αλλά την ε, κυβερνοασφάλεια που αποτελεί πυλώνα της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Κάτι άλλο. Η ευαισθητοποίηση των, σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές δυνατότητες που υπάρχουν. Υπάρχει έλλειψη γνώσεων σε ό,τι αφορά διαφόρων ειδών δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι οι δράσεις θα πρέπει να βασίζονται βάσει στις, ε, μάλλον θα πρέπει να στις ανάγκες και στη ζήτηση που υπάρχει. Αλλά αυτό που θα πρέπει επίσης να λεφθεί υπόψη είναι η μείωση του δημοσίου ελλείμματος και η μείωση του κόστους είναι βασικό ζήτημα στην τρέχουσα φάση. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι οι διαλειτουργικές λύσεις να μην δημιουργούνται από το μηδέν. Ε, υπάρχουν ήδη διαλειτουργικές ε, λύσεις που αναπτύσσονται από διάφορα κρατημέλη στην ε, Φιλανδία, στην Εστονία για παράδειγμα χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα και έτσι γίνεται ανταλλαγή απόψε, πληροφοριών για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα. Είναι λοιπόν σημαντικό να αυξηθεί και η συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία τυποποίησης προκειμένου να είναι πιο σωστό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος, ο κύριος Χέγκελ που αντικαθιστά τον κύριο Τορσανόφσκι, σκιώδη εισηγητή του ECR. Ναι. Ο κύριος Τοζανόφσκι πρέπει να είναι στην πατρίδα του σήμερα και γι' αυτό εγώ τον ε, παίρνω τη θέση του. Κύριε Πρόεδρε, πριν από 20 χρόνια ήμουν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του IBM Europe και πήγα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ζήτησα να κάνει αυτό που κάνουμε σήμερα. 20 χρόνια τη πήρε. Να πω λοιπόν να ευθύ αμέσω ότι βεβαίω είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία αυτή. Είναι μια πρόταση που πραγματικά έπρεπε να είχε ε, λάβει σάρκα και οστά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από την άλλη πλευρά Απογοητεύει το γεγονός ότι μόνο 16 χώρες θα συμμετάσχουν τελικά από ό,τι φαίνεται. Ίσως δεν διαβουλευτήκαμε αρκετά με ορισμένους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτή είναι η πρώτη μου ανησυχία λοιπόν, ότι 16 χώρες μέλη φαίνεται να θέλουν να συμμετάσχουν. Δεύτερη μου ανησυχία είναι η εξή. Πράγματι είναι πολύ καλή πρωτοβουλία, χρειάστηκε 20 χρόνια για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε ότι οι χώρες μας, οι επιχειρήσεις μας, οι ενώσεις μας ανταγωνίζονται τον υπόλοιπο κόσμο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Κίνα, την Ινδία. Και άρα αυτό που λείπει σε όλη την έκθεση είναι ε, κάποιες παραδοχές για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Καλό είναι βεβαίως το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις έχουν ένα αρκετά τυποποιημένο τρόπο για να αντιμετωπίζουν τις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική κτλ. Θα πρέπει όμως να το έχουν αυτό και σε σχέση με τον υπόλοιπο ε, κόσμο, ειδικά με την διευρυμένη κοινή αγορά με το TNP και το CETA. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μαραγκάλ έχει το λόγο σκιώδης εισηγητής ε, για τους πράσινους. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Με ενθουσιάζει η δυνατότητα που έχω να δουλέψω με αυτό το φάκελο. Είναι ένα πεδίο με το οποίο είχα ασχοληθεί για πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πολύ καιρό Βέβαια, όταν εργαζόμαστε στη δημόσια διοίκηση της δικής μου περιφέρειας, της δικής μου χώρας, Κατανοώ και συμφωνώ απολύτως με το πνεύμα της έκθεσης και με τους στόχους που θέτει εκείνη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία, να έχουμε περισσότερες απαιτήσεις από τους εαυτούς μας. Δηλαδή, δεν υπάρχει πρόβλημα με την οπτική γωνία, Συμφωνώ απολύτως με την οπτική γωνία που υιοθετεί η έκθεση. Θέλω όμως να έχει μεγαλύτερη ένταση η προσέγγιση μας. 130 εκατομμύρια μέχρι το 2020 μπορεί να φαίνονται πολλά χρήματα, αλλά δεν είναι και τόσα πολλά τελικά και δεν θα πρέπει ε, να μείνουμε από καύσιμα στη μέση του δρόμου. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος ορίζοντας για το ίσα 2 είναι αρκετά φιλόδοξος και θα είναι ακόμα πιο φιλόδοξο αν μπορούμε να εντοπίσουμε συγκεκριμένους στόχους που δεν αναφέρονται ρητός στην έκθεση σε κάποιους από τους προαναφερόμενου τομείς. Αναφέρθηκαν τα τελωνία, μιλούμε για την κινητικότητα και για τα logistics, τη μεταφορά των εμπορευμάτων, στην πολιτιστική κληρονομιά και σε ορισμένα πεδία των εργασιακών σχέσεων, τη αγορά εργασία έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και υπάρχουν και τα οικονομικά ζητήματα. Ε, π.χ. φορολογική διαχείριση. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διαλειτουργικότητα στην φορολογική διοίκηση. Καλό θα ήταν να Υπάρχουν όλα αυτά και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης και σε επίπεδο ε, δικαστικής διαρρύθμισης. Είναι καλό βεβαίως ότι γίνονται προσπάθειες για μια ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή πέραν των άλλων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη μαύρη οικονομία και να καταφέρουμε να έχουμε σαφή και καθαρά αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και να έχουμε υπόψη μας την τεράστια διαφορά που έχουν οι διάφορες χώρες. Δηλαδή η κάθε μία ξεκινάει από πολύ διαφορετικό σημείο εκκίνησης και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Θα πρέπει κατά ένα μέρος του προγράμματος να γίνεται δουλειά στη σύγκληση έτσι ώστε όλοι να φτάσουν σε ένα περίπου συγκρίσιμο επίπεδο για να μπορέσουν όλοι να αξιοποιήσουν όσο δυνατόν περισσότερο αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό το πρόγραμμα σύγκλησης θα πρέπει να λειτουργήσει υπέρ της ενίσχυσης της εσωτερικής διαλειτουργικότητας στις εκάστοτε χώρες, έτσι ώστε στο εσωτερικό κάθε χώρας να υπάρχει μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, να καλυφθούν νομικά κενά και παραθυράκια. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε τον κύριο Μαρακάλ. Επόμενος ομιλητής θα είναι η κυρία Πιλάρ Δεκαστήγιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ε, μοιραστώ μαζί σας κάποιους προβληματισμούς οι οποίοι αποτελούν και την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτής της έκθεσης. Συμφωνώ βεβαίως με τους στόχους της έκθεσης, ωστόσο η δημόσια διοίκηση έχει ένα τεράστιο ρόλο να διαδραματίσει για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και αυτό συμβαίνει πολύ περισσότερο στη δική μας ε, Ήπειρο από ότι σε άλλες υπήρους και σε άλλες πολιτικές και ε, ένομες τάξεις. Θα πρέπει λοιπόν η δημόσια διοίκηση να λειτουργήσει ως επιταχυντής της ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας. Και γι' αυτό το θέμα της διαλειτουργικότητας είναι ε, εξαιρετικά σημαντικό γιατί έχει αντίκτυπο σε διάφορους παραγωγικούς κλάδους και σε άλλους τομείς που επηρεάζουν άμεσα την πραγματική οικονομία. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ξεκινήσουμε την ομοπαρασκευαστική δραστηριότητα του νέου Κοινοβουλίου και ε, τη δουλειά ε, της Επιτροπής μας. Θέλω λοιπόν να πείσω τους πάντες για το πόσο επίγον είναι όλο αυτό που θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Ε, ε, πόσο επίγουσα είναι η δράση που καλούμαστε να αναλάβουμε στην επόμενη νομοθετική ε, περίοδο, στην επόμενη νομοθετική θητεία ουσιαστικά ε, για να πω μια μεταφορά ε, είναι το last minute call. Είναι σαν να, μας, ε, σαν ήμασταν επιβάτες και να μας φωνάζουν στην πύλη επιφύβασης το τελευταίο λεπτό πριν κλείσουν οι πόρτες του αεροπλάνου. Σε αυτή τη θέση βρισκόμαστε για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτό το αεροπλάνο. Λένε οι συνάδελφοι, είπε ο προηγούμενος συνάδελφος, ότι πριν από 20 χρόνια το ζήτησε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 20 χρόνια έχουν περάσει. Έχω κουραστεί να επαναλάβω τον εαυτό μου. Να επαναλαμβάνω συνεχώς τον εαυτό μου. Ότι έχουμε μια αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών. Είμαστε η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Μπλα μπλα Και, λοιπά και, λοιπά και, και είμαστε, έχουμε μια ενιαία αγορά. Και έχουμε στην περίπτωσή μας την ενιαία ψηφιακή αγορά και με αυτό θα κάνουμε ένα τεράστιο βήμα Ιδαλλιώς θα συνεχίσει η γη να γυρίζει, θα συνεχίσουν οι επιχειρήσεις να παράγουν και οι επαγγελματίες να προχωρούν καλός, αλλά δυστυχώς η ενιαία αγορά δεν θα λειτουργήσει ως επιταχυντής. Εάν δεν πράξουμε, εάν δεν δράσουμε, πραγματικά είμαστε στο παραπέντε. Και αν όχι στο παραπέντε να πω ότι είμαστε στο παραένα. Και πρέπει ως Κοινοβούλιο να το έχουμε υπόψη μας και η Επιτροπή να το έχει αυτό υπόψη της και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε την Πιλάρ, την κυρία Ντεκαστίγιο Λομπελάρ, γιατί εσείς είστε άλλωστε η βασική μας εισηγήτρια στον τριμερή διάλογο για την ψηφιακή ατζέντα και την αγορά τηλεπικοινωνιών. Και ελπίζουμε ότι ο τριμερής διάλογος να ξεκινήσει ως να τον νωρίτερα. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσει το Δεκέμβριο. Ζήτησα από την Ιταλική Προεδρία να ε, προχωρήσει το θέμα. Και η Ιταλική Προεδρία υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος τον Δεκέμβριο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και θα είναι πολύ καλό να ε, έχουμε το εναρκτήριο λάκτισμα του διαλόγου το Δεκέμβριο. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ταμπουράνο, που θα αντικαταστήσει τον κύριο Μπορέλη Σκιώδη εισηγητή από το EFTD. Κύριε Ταμπουράνα, παρακαλώ. Χαίρετε Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους τους συνάδελφους εκ μέρους, συναδελφούς, εκ μέρους του κυρίου Μπορέλη και ο οποίος ζητά συγγνώμη για την απουσία του γιατί πρέπει να παραστεί την διασκέδευση των Προέδρων να σας μεταβιβάσω τα εξής για την διαφωνία αρμοδιοτήτων που πρέκυψε μεταξύ της Επιτροπής μας και της ΕΜΚΟ. Παρόλα αυτά όλοι συμφωνούμε για τη μεγαλύτερη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μας και την διαλειτουργικότητα των επιγραμμικών υπηρεσιών, ιδίως για τα κάτι μέλη που πρέπει να ανακτήσουν σε αυτό το τομέα. Οι υπηρεσίε όπω οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί, οι ηλεκτρονικέ δημόσιε προμήθειε και η ηλεκτρονική υγεία είναι θέματα που δεν μπορεί παρά να αυξήσουν την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρει ο δημόσιο τομέα στου Ευρωπαίου πολίτε. Από την πλευρά μα λοιπόν είμαστε στη διάθεση συνεργασία, σε πλήρη προθυμία συνεργασία για το θέμα αυτό παρά την ε, σύντομη λήξη προθεσμία ε, ε υποβολή τροπολογιών το Δεκέμβριο του 2015. Να προσθέσω στη, τη δική μου σύντομη συμβολή ότι θα πρέπει να κάνουμε το δυνατόν περισσότερο για να να εγκριθούν λειτουργικέ πλατφόρμες με συστήματα όχι αποκλειστική ιδιοκτησία, και με το σύστημα των προγραμμάτων Open και ISO. Ε, και αυτά τα έχει ήδη το ίδιο κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν εμείς οι ίδιοι να αρχίσουμε να δίνουμε το σωστό παράδειγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω να ζητά άλλος κανείς το λόγο. Οπότε, να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μαργαρίτα Αλμπερκάσης, να τοποθετηθεί για αυτό το θέμα, εάν μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τη γενική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σταθώ σε μερικά από τα σημεία που έφυξαν οι διάφοροι ομιλητές Το πρώτο που σημείωσα, πολύ σημαντικό θέμα, καλύπτεται από το νέο πρόγραμμα και τη νέα μορφή του προγράμματος το Connecting Euro Facility, ο μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη. Όπως βλέπετε, στην πρόταση στοχεύουμε στη διαλειτουργικότητα και λύσεις για συνεργασία δημόσιων διοικήσεων μεταξύ τους στην Ευρώπη αλλά και τη σχέση τους με τους πολίτες. Έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση. Η οριζόντια δεν σημαίνει ότι θα βρει όλες τις λύσεις μόνη της και ότι θα προσφέρει όλες τις λύσεις διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη. Στην κάθε στον κάθε τομέα ε, υπάρχει μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις ξεχωριστά. Το πρόβλημα που έχουμε σήμερα δεν αντιμετωπίζονται οριζοντίως οι λύσεις που προσφέρονται. Ο καθένας ε, ε, εντοπίζεται στην, στις υποδομές ή στο format ή στην στο περιεχόμενο, εδώ πρέπει να καλύψουμε αυτό το χάσμα και να στηρίξουμε άλλε πρωτοβουλίε. Λόγω χάρη στο πλαίσιο τη πρωτοβουλία για τη διασύνδεση τη Ευρώπη και στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων, στον τομέα τη κοινοτομία και τη έρευνα, για παράδειγμα, πρέπει να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ των λύσεων που ήδη έχουν ε, βρεθεί μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και των λύσεων που θα αρχίσουν να λειτουργούν στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για την διασύνδεση της Ευρώπης. Το ανέφερε και ένας βουλευτής εδώ, τον, ε, το σύστημα αυτόματης μετάφρασης και τις υπηρεσίες αυτόματης μετάφρασης. Ε, το EASY το έχει ήδη προσφέρει αυτό και θα το αναλάβει ως υπηρεσία το διασυνδέοντας την Ευρώπη. Θα μπορέσουν έτσι να το αξιοποιήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Όμως από την άλλη, όπως το Άιζα σήμερα, θα πρέπει οι λύσεις αυτές να διαδοθούν και στο μέλλον. Η λύση λοιπόν αυτή της αυτόματης μετάφρασης θα διατεθεί από τις ε, δημόσιε υπηρεσίε που ήδη τη διαθέτουν προς τις άλλες, θα την πάρουν από την κοινή πλατφόρμα και θα τα εφαρμόσουν στη δική τους μηχανή. Θα χρησιμοποιηθεί λοιπόν ως υπηρεσία από το σύνολο των λύσεων που προσφέρεται ή ως λύση μεταξύ των λύσεων που θα διτεθούν στις δημόσιες δικήσεις. Αυτή είναι μια ενδεχόμενη σχέση του Άιζα με τα υπόλοιπα προγράμματα. Ένα άλλο σχόλιο που άκουσα είναι τα πρώτα βήματα που μπορεί να κάνει και να προβλεφθούν για το ΆΙΖΑ 2. Προτείνονται διαφορετικές λύσεις από όσα έχει προβλέψει το οικοδόμημα για την ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα και τη σχετικό χάρτη. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια τέλεια χαρτογράφηση του τι υπάρχει στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στις δικήσεις των κρατών μελών. Ιδάλλως δεν γίνεται να δούμε πού θα πρέπει να εντοπίσουμε τις προσπάθειές μας. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η χαρτογράφηση των υπερχουσών λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε, στις εθνικές διοικήσεις. Όπως πολύ σωστά υπόθηκε, οι δημόσιες διοικήσεις έχουν ε, ήδη προβλέψει κάποιες λύσεις που άλλες χώρες δεν τις διαθέτουν και θα μπορούσαν να τις αξιοποιήσουν. Όμως προηγουμένως πρέπει να το μάθουν. Πρέπει λοιπόν αυτά να διατεθούν, να διαδοθούν, να μπορεί κανείς να κάνει αναζήτηση σε αυτά τα πεδία και με απλό τρόπο. Αυτό είναι ο ρόλος της πλατφόρμας. Και για να φτάσω και στο συμπέρασμα της παρέμβασής μου, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μόνο 16 χωρών ε, στην πρόταση για το ΆΙΖΑ, έχουμε υπόψη ότι θα γίνουν πολλές αξιολογήσεις εδώ. Η πρώτη αφορούσε τη στρατηγική την ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Διαλειτουργικότητας και την ε, ε, επισκόπησή της και την αξιολόγηση. Και υπάρχει και το παρατηρητήριο για τη διαλειτουργικότητα που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες διαλειτουργικότητας από όλα τα κράτη-μέλη και φροντίζει να τις μεταδώσει. Το άλλο στοιχείο ήταν η ενδιάμεση αναθεωρήση του προγράμματος ΆΙΖΑ που ήδη έγινε και επίσης τα αποτελέσματά της διαδόθηκαν παντού και είχαν πλήρη συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια των διαβουλεύσεων οι εκπρόσωποι των κρατών μελών με την αρμόδια επιτροπή, με τη συμμετοχή όλων για να ελέγξουν την πρόταση ΆΙΖΑ που έχετε τώρα στο τραπέζι σας, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Να ζητήσω από τον εισηγητή μας, τον κύριο Κάρλος Ζωρίνιου, να ε, δώσει τέλος τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τους άλλους συναδέλφους για τις συνεισφορές τους. Από τη συζήτηση αυτή καταλαβαίνω ότι οι επτά τομείς που εντόπισα ως τομείς όπου θα μπορούσαμε να πετύχουμε μικρές βελτιώσεις, την χάνουν γενικές αποδοχές. Και συμπεραίνω ότι θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο έντονοι στις εκφράσεις μας σε κάποιες ε, περιοχές. Ως προς τις προθεσμίες, το timing, την κατεπίγουσα ανάγκη κάποια θέματα να προωθηθούν, Πρέπει το πρόγραμμα αυτό δηλαδή να είναι πλήρως λειτουργικό από 1η Ιανουαρίου 2016, αλλά πρέπει να είναι και επικαιροποιημένο, δηλαδή να είναι λειτουργικό ακριβώς με τις τεχνολογικές εξελίξεις, με τις ε, διαφορές και τα όσα έχουν προκύψει ως, ε, την 1η Ιανουαρίου 2016. Τώρα, ως προς το συγχρονισμό μεταξύ προγραμμάτων, Α είναι σαφέ ότι απόφαση και να πάρουμε, ότι το ΙΖΑ 2 θέλει να δημιουργήσει μια ε, πλατφόρμα, μια οριζόντια πλατφόρμα συνεργασία για τις 28 χώρε. Όμως, έχοντας χάσμα, ψηφιακό χάσμα μεταξύ διαφόρων χωρών, είπε ο κύριος Μαραγκάλ έναν τρόπο να καλυφθεί το ε, χάσμα που ήδη υπάρχει με τη σύγκληση. Άλλος τρόπος είναι να διευκολύνουμε και να δώσουμε κίνητρα για να βρεθούν λύσεις διακρατικές. Χώρες με μικρότερες ή μεγαλύτερες ψηφιακές δυνατότητες. Αυτή η μεγαλυτερες ψηφιακες δυνατοτητες αυτη κοινή αντιμετώπιση των αναγκών μπορεί να οδηγήσει στην πραγματική βελτίωση. Επίσης θα μπορούσε να υπάρχει ένα πρόγραμμα εντατικής ε, ενημέρωσης για την απόφαση αυτή, να την ε, γνωρίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, να είναι ευρέως γνωστή, να, είναι, να μην είναι απλώς μια τεχνοκρατική απόφαση, αλλά μια απόφαση τεχνοκρατική που θα συμβάλλει τελικά στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Θα μπορούσαμε λοιπόν μέρος των κονδυλίων που προβλέπονται να τα αφιερώσουμε στην ε, προβολή των λύσεων που προτείνουμε. Και για μια ερώτηση που τέθηκε εδώ, η οποία είναι αρκετά δύσκολη, ένα θέμα περίπλοκο. Μιλάμε για τη λειτουργικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά ταυτόχρονα συζητάμε τη συμφωνία TTIP, μετά τη συμφωνία με τον Καναδά και άλλες ασιατικές χώρες. Εδώ πώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε την διαλειτουργικότητα και με άλλα μέρη του κόσμου. Αυτά είναι τα συμπεράσματα της δουλειάς μας που ελπίζω να προχωρήσει γρήγορα από εδώ και μπρος, Πρόεδρε. Από το Σεπτέμβριο περιμένουμε η έκθεση αυτή να ε, προχωρήσει. Ξέρετε ότι δεν έχει αποπλέψει ακόμα η πρόταση αυτή. Βέβαια ο εισηγητής έχει ξεκινήσει τη δουλειά του, αλλά ξέρετε ότι περιμένουμε να προχωρήσει ακόμη πιο γρήγορα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκα, θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Έχω δύο παρατηρήσεις να κάνω. Καταρχάς πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι λίγο δειλή, σαν να πρέπει να την ενθαρρύνουμε περισσότερο για τις προτεραιότητες αυτές, ε, για να έχει χρονοδιάγραμμα. Και για να έχουμε χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ βασικά πράγματα και σοβαρά πράγματα. Από τα πιο αρνητικά, από τα πιο δύσκολα, τα πιο δυσεπίλητα. Για παράδειγμα η φορολογική διοίκηση. Κάθε χρόνο χάνουμε 300 εκατομμύρια ευρώ λόγω της ανικανότητας της διοίκησης και η κλασική διαλειτουργικότητα υπάρχει, θα μπορούσε να γεμίσει το κρατικό κορβανά, θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων διοικήσεων. Υπάρχει αυτή η λύση και δεν υλοποιείται. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαλέξει την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Καλό πράγμα είναι η, αυτόματη μετάφραση, αλλά καλύτερο είναι να έχουμε καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών εν μέσω μεταξύ φορολογικών διοικήσεων. Γιατί φορολογικές διοικήσεις έχουν εργαλεία πληροφορικής με πολύ καλές επιδόσεις, αλλά δεν διαδίδουν τις πληροφορίες αυτές. Τα τελωνία, για παράδειγμα, οι άλλες υπηρεσίες έχουν εξαιρετικά συστήματα πληροφορικής και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Μπορούμε λοιπόν να υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση, να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και ο εισηγητής μας λοιπόν, ο συνάδελφος Ζωρένιο, θα προετοιμάσει το σχέδιο έκθεσης του θα εξετάσουμε το σχέδιο της έκθεσης στις 22 Ιανουαρίου 2015. Ακρόαση για το ΙΖΑ 2. 22 Ιανουαρίου επίσης. Προθεσμία για τα κατάθεση τροπολογιών. Έξι μέρες αργότερα, στις 28 Ιανουαρίου 2015, στις 12 το μεσημέρι. Ψηφοφορία στην Ήτρε. 14 Απριλίου 2015. Και μετά τον Ιούνιο στο 2015. Αυτό είναι το προκαταρτικό μας χρονοδιάγραμμα. Και ο εισηγητής είναι υπεύθυνο για όλες τις φάσεις. Μπορείτε να μου έχετε πιστοσύνη, Πρόεδρε θα τα κάνω όλα όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για τη συζήτηση αυτή, για την δραστηριότητά σας και τον συνάδελφο Νίκα για τις παρατηρήσεις που έκανε, πάρα πολύ σημαντικές και αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια. Και αυτό πολύ σημαντικό ζήτημα. Να σας επενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια το Μάιο του τρέχοντος έτους, μετά την ε, κρίση στην Ουκρανία. Πλέον είναι ακόμα πιο κατεπήγον το ζήτημα. Είμαστε στα πρότρια του χειμώνα. Η Ήτρε αποφάσισε να καταρτήσει έκθεση πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια. Και κάναμε και ακρόαση σχετικά στις 5 Νοεμβρίου. Ανταλλαγή λοιπόν απόψε για πρώτη φορά σήμερα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, το θέμα αυτό, παρομοίως όπως και στο σημείο 5, για τις λύσεις διαλειτουργικότητας. Η συζήτηση αυτή γίνεται πριν από το σχέδιο της έκθεσης. Να καλέσω τον κύριο Σαντάργας να παρουσιάσει την άποψή του, τις θέσεις του. θα συμπεριληφθούν ασφαλώς στο σχέδιο έκθεσης που θα παρουσιαστεί στην συνεδρίαση της Ήτρε τον Γενάρη που θα είναι γεμάτη, πληρέστατη. Σας δίνει το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως αναφέρατε ήδη, η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει. Γίνονται και σημαντικές ε, συνεδριάσεις, γύρι τραπέζις για διάφορα ζητήματα. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν πολύ εμπεριστατωμένη όσο πιο πολλές πτυχές γινόταν της ενεργειακής ασφάλειας αλλά θέλαμε να επιλέξουμε τα πιο σημαντικά ζητήματα για την έκθεση. Η έκθεση δε θα είναι έτοιμη, Ένα το χρόνο, την άλλη εβδομάδα. Να ευχαριστήσω τους κοιόντες συζητητές. Έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων τις ιδέες τους να τις ενσωματώσω και αυτές μέσα στην έκθεση. Όπως ανέφερα, η ανακοίνωση είναι περιεκτικότατη, σύνθετη. Άρα, θα κάνω κάποια γενικά σχόλια. Στην έκθεση γενικά αποφασίσαμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης της ενεργειακής ασφάλειας, γιατί είναι ξεχωριστά πράγματα. Και στην αρχή κάναμε κάποιες εισαγωγικές ε, παρατηρήσεις. Φυσικά, ο βασικός λόγος, ίσως και ο μόνος λόγος άλλωστε της συζήτησης, είναι τα προβλήματα εισαγωγών αερίου μέσω της Ουκρανίας και ο επερχόμενος χειμώνας. Στην έκθεση αυτή, ωστόσο, πιστεύουμε, όπως και να έχει, θα ψηφιστεί μετά το χειμώνα. Άρα δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στα βραχυπρόθεσμα ζητήματα. σε αυτά που αποφασίστηκαν να γίνουν, stress test και ούτω καθεξής, αλλά κοιτάμε και την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διάσταση βασικός στόχος είναι η ενεργειακή ένωση ασφαλώς, προκειμένου η ενεργειακή ασφάλεια να καταστεί πραγματικός πυλώνας μαζί με την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα της ενέργειας στο μέλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό. Η εσωτερική διάσταση εμπεριέχει ασφαλώς και είναι λογικό τα θέματα ζήτησης σε ό,τι αφορά την ενέργεια φυσικά καταρχάς μέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας. Προφανώ αναφέρουμε και την ε, οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα, για την ε, εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και καλούμε να εφαρμοστούν όλες οι σχετικές διατάξεις. Επόμενο σημαντικό στοιχείο είναι η εγχώρια παραγωγή ενέργειας. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η εγχώρια παραγωγή ενέργειας θα πρέπει να καλύπτει όλη την αλυσίδα της παραγωγής ενέργειας. Όχι μόνο δηλαδή η πηγή ενέργειας να είναι χώρια, αλλά και η τεχνολογία, οι εγκαταστάσεις να είναι ευρωπαϊκές. αυτά λοιπόν για την εσωτερική ευρωπαϊκή παραγωγή ενέργειας. Αυτό καλύπτει ασφαλώς κατά κάποιο τρόπο αυτά που αναφέρονται στην τεχνολογία της ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ να είμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενεργειακή αγορά, ενοποιημένη ενεργειακή αγορά, φυσικά αποσκοπεί στην ενεργειακή ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και διασυνδέσεις, υποδομές, MPCIs. Θα πρέπει όλα αυτά να εφαρμόζονται το συντομότερο δυνατό. Η εξωτερική τώρα διάσταση. Σαφής και αυτή θεωρώ, αλλά επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω κάποιες πτυχές. Καταρχάς, μία πηγή εφοδιασμού. Αυτό είναι μια σημαντική διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση όμως αυτή είναι τόσο σημαντική που σημαίνει ότι θα πρέπει να κινηθούμε και προς αξιόπιστες πηγές. Και θα κλείσω λέγοντας το εξής. Αυτό που είπα και στην αρχή. Μάθαμε πρόσφατα η Ρωσία δεν αποτελεί πλέον αξιόπιστο πάροχο. Αυτό υπογραμμίζεται ξεκάθαρα γιατί ρήτα αρνούνται να συμμορφωθούν με το ευρωπαϊκό δικτύο. Δίκαιο. Και η ενεργειακή παροχή είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούν επανειλημμένα και συστηματικά ως πολιτικό εργαλείο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Τώρα εισηγητή, εισηγητές. Ο κύριος Πόχε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σωστά τα λέτε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακοίνωσή της. Καλωσορίζω την ανακοίνωση αυτή, η οποία διατυπώθηκε τον Μάιο, και το λέω αυτό διότι η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγωγές είναι οικονομικό ζήτημα, οικονομικό πρόβλημα, αλλά και πολιτικό πρόβλημα για τις περισσότερες χώρες. Χρειάζεται λοιπόν δράση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε τους πόρους, πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη και να διαχειριστούμε τη ζήτηση καλύτερα. Δύο είναι αυτά τα οποία θα ήθελα να αναφέρω και πιο συγκεκριμένα μάλιστα. Πρώτον, η επάρκεια της ενέργειας δεν θα πρέπει να ορίζεται μόνο από την τιμή και τη διαθεσιμότητα, αλλά και από την αηφορία και τη σταθερότητα του συστήματος συνολικά. Πρέπει να ορίζεται αυτό το σύστημα έτσι ώστε να καταπολεμά την ενεργειακή φτώχεια που υπάρχει σε ορισμένα κράτη-μέλη. Έρχομαι τώρα στο όραμα. Η σημερινή κατάσταση μπορεί να γίνει ανεκτή μόνο σε μεσοπρόθεσμη βάση. Πρέπει να το δούμε το θέμα πιο μακροπρόθεσμα, να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Και αυτό είναι κάτι που συζητήσαμε και με τους υπολείπους ε, σκιώδεις εισηγητές. Ήταν μια πολύ παραγωγική συζήτηση και σας ευχαριστώ για αυτή. Η στρατηγική λοιπόν για την ενεργειακή επάρκεια ε, και ασφάλεια θα πρέπει να μην είναι μόνο μεσοπρόθεσμης βάσης, θα πρέπει να εξετάζει και την αξιοπιστία των υφιστάμενων συστημάτων. Και θα ήθελα να τονίσω και κάποια πράγματα που νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν στην έκθεση. Πρώτον, η επένδυση στην τεχνολογία, τεχνολογία που θα μας επιτρέψει να εξυγχρονίσουμε το ενεργειακό μείγμα σε κάθε κράτος μέλος. Ε, παραμένοντας όμως τεχνολογικά ουδέτεροι, για να μπορεί το κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει το ίδιο πώς θα αξιοποιεί την ενέργειά του και από πού θα βρίσκει τις πηγές ενέργειάς του αναλόγως με τους δικούς του στόχους και σκοπούς. Ενεργειακή αποδοτικότητα, ενεργειακή εξοικονόμηση, ενεργειακή ασφάλεια, επάρκεια, όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε σε πιο βραχυπρόθεσμη βάση και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έτσι τη ζήτηση. Είναι θέμα υποδομών. Ε, υπάρχουν ας πούμε project, υπάρχουν έργα κοινού ενδιαφέροντος, κοινού συμφέροντος. Πρέπει να έχουμε την έξυπνη σύνδεση στο σύστημα. Το smart grid, η έξυπνη σύνδεση ε, σύστημα θα είναι ο τρόπος και η λύση να ανταποκριθούμε στις υψηλές διακυμάνσεις των τιμών, στις υψηλές διαφορές μεταξύ προσφοράς, ζήτησης και το καθεξής. Μία ενεργειακή αγορά που λειτουργεί. Εάν την πετύχουμε, δεν θα εξαρτώμαστε τόσο από προσφορά που να διακυμαίνεται και να κυμαίνεται και να αποκατεβαίνει από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτά πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ashley Fox από το ECR, Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Σάουνταργκας γιατί μοιράστηκε μαζί μας τις αρχικές του για το φάκελο αυτό στη συνάντηση με τους κοιόδιους συζητητές την περασμένη εβδομάδα. Ήταν πολύ χρήσιμη η συνάντηση και τον ευχαριστώ για αυτή. Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη είναι ζωτική σημασία για την ευμερία ε, των οικονομιών των κρατών μελών και κλειδί για την επίτευξη αυτή τη ασφάλεια είναι μια πλήρω λειτουργούσα ενιαία αγορά με διαλειτουργικότητα έτσι ώστε η παροχή, η προσφορά να κιλά, απρόσκοπτα σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε διαφοροποιημένε πηγέ προμήθευσης για να αντιμετωπίζουμε τον ανταγωνισμό. Πρέπει να έχουμε σαφείς στόχους, να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να αποφασίσει το καθένα ποιο είναι το καλύτερο ενεργειακό μείγμα για το ίδιο. Συμφωνώ με τον κύριο Σάουντοργκας. Αν αυξήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα και μετριάσουμε τη ζήτηση, τότε θα είμαστε σε ε, καλύτερη θέση. Πρέπει να στηρίξουμε τις καινοτόμε τεχνολογίες που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε αυτό το σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, μία ενιαία αγορά μία και μόνη, ευρύθμως λειτουργούσα, η οποία θα δίνει στα κράτη-μέλη την ασφάλεια που χρειάζονται. Αυτό είναι το βασικό. Ξέρετε, μεγάλο μέρος της ολοκλήρωσης της ενεργειακής αγοράς μέχρι σήμερα ε, λαμβάνει χώρα στη Βόρεια και στη Δυτική Ευρώπη. Ε, αν δεν γίνουν διασυνδέσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο που μας αφορά, στο κομμάτι που γεωγραφικά αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα ε, προχωρήσουμε επαρκώς. Μιλούμε για παράδειγμα την κατάσταση μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Οι επτά σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ισπανίας έχουν το δυναμικό να τροφοδοτήσουν όλη την Ευρώπη. Ωστόσο η Γαλλία είναι επιφυλακτική και δεν θέλει να επιτρέψει στο έδαφος της έναν διασυνδετή τι, να το πω έτσι, interconnector, ένα ε, συνδετικό κρίκο μεταξύ των 7 τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ισπανίας και την υπόλοιπη Ευρώπη. Τι θα κάναμε με την Ουκρανία, είδατε τι έγινε, πώς θα μπορούσαμε να έχουμε αντικαταστήσει ε, τις ε, ρωσικές εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είχαμε το λειτουργικούς τους 7 τερματικούς σταθμούς της Ισπανίας, δεν θα μας ενδιαφέρει αν ο κύριος Πούτιν ε, κλείσει ή έκλεινε τη στρόφιγγα. Καθόλου μάλιστα. Και αυτό είναι σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επενδύσουμε σε βασικά project υποδομής, να δίνουμε προτεραιότητα σε όλα αυτά τα έργα που είναι κρίσιμη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Πρέπει να δώσουμε σε όλα αυτά την απαραίτητη και πολιτική αλλά και οικονομική στήριξη και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το τρίτο ενεργειακό πακέτο υλοποιείται πλήρως από όλα τα κράτη-μέλη θα ανοίξουν έτσι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, θα επωφεληθούν οι καταναλωτές από αυξημένο ανταγωνισμό και άρα χαμηλότερες τιμές. Σε κάθε περίπτωση κατά την αγορά τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα κατά την αγορά την προμήθευση να επιλέξουν αυτό που νομίζουν και αυτό που επιθυμούν. Δεν θα πρέπει να έχουμε συλλογικές συμφωνίες προμήθευσης από πάνω προς τα κάτω τις οποίες να καθοδηγεί, η Ευρωπαϊκή, να καθοδηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αυτό θα διαστρεβλώσει την αγορά. Η αγορά είναι το κλειδί για την ενεργειακή επάρκεια, για την ενεργειακή ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει βήματα για να βοηθήσει την κατάσταση, μετά όμως θα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της ότι δεν χρειάζεται πια η παρουσία της να αποσυρθεί και να αφήσει την αγορά να ρυθμιστεί και να λειτουργήσει. Στη δική μου χώρα, ξέρετε, Έχουμε έναν ηγέτη εργατικών αρκετά ανόητο που υποσχέται ότι θα παγώσει τις τιμές για 12 μήνες. Δημιουργεί ανασφάλεια στις επιχειρήσεις, χαμηλότερες επενδύσεις και άρα υψηλότερες τιμές στους καταναλωτές σε βάθος χρόνου μετά το πέρας των 12 μηνών. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος, κύριος Μόρτον Χάλβεκ Πέτελσεν, εκ μέρους των Φιλελεύθερων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική συνεργασία για το θέμα αυτό και τους υπόλοιπους συναδέλφους για τη σαφή προθυμία να βρούμε τόπο για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Όλα νομίζω ότι αναγνωρίζουμε την πρόκληση που πολλές ευρωπαϊκές χώρες ε, αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια του εφοδιασμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα θέρμανσης στην καρδιά του χειμώνα που συχνά είναι θέμα ζωής και θανάτου. Η χώρα μου, η Δανία, αντιμετώπισε τη δεκαετία του 70 μια κρίση της ενέργειας που ε, τη λύσαμε κλείνοντας τα φώτα και θέρμανση. Τότε λοιπόν είχαμε αποφασίσει, αποφασίσαμε να μην παραμείνουμε εξαρτημένοι από τον ενεργειακό αφοδιασμό, αλλά να καταστούμε ανεξάρτητοι μειώνοντας την χρήση ενέργειας μέσω της αποτελεσματικότητας και χρησιμοποιώντας ε, ό,τι μέσο είχαμε στη διάθεσή μας ε, και την, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιομάζα κτλ. Θυμάμαι συζητήσεις στη δεκαετία του 70 όπως για παράδειγμα την απαγόρευση χρήσης αυτοκινήτων τις Κυριακές προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να μειωθεί η κατανάλωση. Πλέον η Ιδανία δεν εξαρτάται τόσο πολύ, δεν εξαρτάται από το πετρέλαιο και από ενεργειακές ε, πηγές και αναδύεται στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε καταδείξει πως είναι δυνατόν να υπάρξει μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να υπάρχει και αποτελεσματικότητα της χρήσης της ενέργειας, αλλά και ανεξαρτησία και οικονομική. Είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να βρούμε τις καλύτερες λύσεις σε ό,τι αφορά και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια ενεργειακή σε όλη την Ευρώπη. Οι χρηματοοικονομικές, ε, οι χρηματοοικονομικοί πόροι που διατύφονται ήδη από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και από τις ε, δημόσιες επενδύσεις, στο πακέτο Juncker όπως ονομάζεται, θα υποστηρίξουν φαντάζομαι προγράμματα που θα συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια και εκ παραλλήλου θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο με μια τόσο συνεκτική και ολιστική προσέγγιση μπορούμε να δώσουμε μια να τονώσουμε την ανάπτυξη και να φροντίσουμε προκειμένου να μην συνεχίσουν οι πολίτες μας να είναι θύματα εκβιασμού σε ό,τι αφορά την ε, παροχή ενέργειας. βλέπω στη στενή συνεργασία με τους Κιώδης και με τον εισηγητή και ανυπομονώ να ακούσω και τη σχετική συζήτηση. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Ο κύριος Ηλικιώτης. Ε, πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο του Σαουτάρκας ε, για τη χρήσιμη συνάντηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα στο Στασβούργο και μας δίνει την ευκαιρία μέσα από μια συλλογική προσπάθεια να ετοιμαστεί από τον ίδιο όσο καλύτερα μια πιο ολοκληρωμένη έκθεση. Ε, κατά την άποψή μα, η της ΓΚΟΕ η ανακοίνωση τη Επιτροπή έχει αρκετά κενά. Ε, για μα, η ανάγκη ενίσχυση τη ενεργειακή ασφάλεια απορρέει πρωτίστω από το γεγονό ότι η ενέργεια σήμερα συνιστά βασικό ανθρώπινο αγαθό, στο οποίο πρέπει να έχουμε όλη πρόσβαση ε, και να έχουμε πρόσβαση, ισότιμη πρόσβαση και ε, σε ευθυνή ενέργεια. Υπάρχουν πολλά να γίνουν προ αυτήν την κατεύθυνση, τα οποία πρέπει να υπογραμμίσουμε και στην έκθεση τη Επιτροπή μα για την ενεργειακή ασφάλεια. Εγώ θα σημειώσω μόνο ε, τρία στοιχεία εδώ. Το πρώτο, τα οποία κατάθεσα και στη συνάντηση που είχαμε με ε, τον εισηγητή και του κοιόδη εισηγητέ. Το πρώτο είναι ότι στι προτεραιότητε μα θα πρέπει να καταγραφεί η ανάγκη να καταπολεμήσουμε την ενεργειακή φτώχεια. Αυτό το νέο φαινόμενο που μαστίζει σήμερα πολλά κράτη και περιοχέ της Ευρώπης. Και ε, χρειάζεται ακριβώς ε, να εντοπίσουμε αυτό το φαινόμενο και να καταθέσουμε εισηγήσει. Το δεύτερο είναι εξίσου σημαντικό να τονίσουμε την άμεση ανάγκη προώθησης μέτρων στο πλαίσιο της ε, ενεργειακής στρατηγικής για άρση της απομόνωσης κρατών ή και περιοχών από τα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα. Δυστυχώς, ενώ εδώ τέθηκε ο στόχος εδώ και πολλά χρόνια, για να τερματιστεί από απομόνωση κρατώ μέχρι το τέλος του 2015 ε, δεν βλέπουμε να υλοποιείται αυτός ο στόχος. Το τρίτο, ε, για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς επιβάλλεται ως Ευρωπαϊκή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα προκειμένου να απεξαρτηθεί από τα ενεργειακά μονοπόλια και να επιτύχει ενεργειακή αυτάρκεια. Επιβάλλεται λοιπόν να αξιοποιήσουμε τις προοπτικές που δημιουργούνται με τα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και ειδικότερα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ενός κράτους μέλους όπως ε, είναι η Κύπρος. Ε, θεωρούμε λοιπόν σημαντικό να υπάρχει στην έκθεση ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την υλοποίηση ενός μεσογειακού κόμβου μέσω διαδρόμου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη καθώς και την πρόταση για χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Ιδιαίτερα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα η νοτιοανατολική Ευρώπη η οποία σήμερα αντιμετωπίζει επίγουσες ανάγκες όπως θεωρούμε και λόγω ακριβώς ε, της, λόγω της ακύρωσης του νότιου διαδρόμου ε, ε, φυσικού αερίου αλλά και των προβλημάτων που υπάρχουν στην Ουκρανία και θεωρούμε ότι από αυτήν την περιοχή μπορεί να ενισχυθεί και ολόκληρη η Νότια Ευρώπη. Ε, και είναι εξίσου σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλίε για την ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα τη ενέργεια με τι χώρε τη Ανατολική Μεσογείου και αναφέρομαι στι τρίτε χώρε πέραν τη Κύπρου που είναι κράτο μέλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Εκ μέρους των Πρασίνων τώρα, ο κύριος Γιάβορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενώσω τη φωνή μου με όσους ευχαρίστησαν την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημοσίευση αυτής της στρατηγικής και τον εισηγητή μας για την πρωτοβουλία να συζητήσουμε και να έχουμε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεσή του από την πλευρά των πρασίνων. Πιστεύω και εγώ ότι είναι σημαντικό για τη στρατηγική να έχουμε αυτόν τον κατάλογο ε, έξι και ενό σημείων. Πολύ σύντομα. Πρέπει να είμαστε πρώτα απ' όλα βέβαια για τη στρατηγική και τη διαδικασία της. Η στρατηγική ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς καμία συζήτηση με το Κοινοβούλιο, με προσώπους της κοινωνίας των πολιτών, βλέπουμε να έχουμε μια πανέτοιμη στρατηγική και πολύ μικρή δυνατότητα να επηρεάσουμε το τελικό αποτέλεσμα, την τελική της μορφή. Αυτό νομίζω ότι εγείρει ερωτήματα περί δημοκρατίας. Ως προς την καρδιά του ζητήματος, έξι είναι οι σημαντικοί τομείς που θα θέλαμε να ενισχυθούν. Πρώτα απ' όλα, η στρατηγική δεν πρέπει να παραμείνει απομονωμένο έγγραφο. Πρέπει να συσχετιστεί με άλλες στρατηγικές και μέτρα της Ένωσης, μεταξύ των οποίων το ενεργειακό πακέτο και η στόχοι για το 2030, η ενεργειακή στρατηγική την Ευρώπη, το σύστημα ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπών και ούτω καθεξής. Πρέπει όμως να υπάρχει και ένα master plan, ένα σφαιρικό στρατηγικό σχέδιο. Τι θέλουμε να πετύχουμε. Ενέργεια με κοινωνικές τιμές, με περιορισμό χρήσης του άνθρακα, Ποια είναι η ουσία της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Η πεποίθηση μου είναι ότι πρέπει να επιδιώξουμε την απαλλαγή εξάρτησης από τον άνθρακα, να παραμένουμε πιστοί στους στόχους της ενεργειακής πολιτικής 2030 και της Ευρώπης 2020 και να μην δεχτούμε οποιαδήποτε αύξηση εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή διοξιδίου του άνθρακα είτε είναι εγχώριες είτε όχι. Δεύτερο σημείο. Η στρατηγική δηλώνει ότι εάν γίνουν όλα όπως τα προβλέπει η στρατηγική, θα αυξηθεί η εξάρτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση από το ρηκτά καύσιμα. Δεν θα μειωθεί, θα αυξηθεί. Οπότε τα μέτρα που περιλαμβάνει η στρατηγική και που επικεντρώνονται στι υποδομέ για το αέριο δεν είναι αρκετά για να μα απαλλάξουν από την ενεργειακή μα εξάρτηση. Θέλουμε λοιπόν και την ενεργειακή αποδοτικότητα για να ελέγχεται η ζήτηση ενέργειας, αλλά θέλουμε και μεγαλύτερη τόνωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έπειτα η ενεργειακή ένδυα. Το θέμα αυτό αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο της ΚΟΕ. Ε, η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι απλώς ασφάλεια της ε, προμήθειας, αλλά και ασφάλεια πρόσβασης. Πρόσβασης του καθενός από τους Ευρωπαίους πολίτες στην ενέργεια. Δεν μιλάμε για μια τεχνητή μείωση των τιμών όμως, αλλά οι πολίτες και τα νοικοκυριά να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια χάρη στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τα σχετικά μέτρα ή τι επενδύσει μας. Αυτό πρέπει να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Τέταρτον, το ενεργειακό σύστημα που θέλουμε να διαμορφώσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε, ε, ε, έχουμε επαναπαυθεί στα ορεκτά καύσιμα και στην πυρηνική ενέργεια. Εάν θέλουμε ενεργειακή αποδοτικότητα, μείωση της ε, ζήτησης ενέργειας και ανθεκτικότερο σύστημα ενέργειας, πρέπει να επενδύσουμε στα ευφυή e δίκτυα, στην, στα αποκεντρωμένα συστήματα. Μόνο έτσι θα πετύχουμε το στόχο μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέμπτον, το δημοσιονομικό σκηνικό. Μπορεί να λέμε ωραία λόγια για την ε, ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα, τα ανανεώσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όμως Εν τέλει, αυτό που πρέπει να απαντήσει που είναι πού θα βρει λεφτά. Μιλάμε για ευρωπαϊκά κονδύλια, πώς θα καταναμηθούν αυτά, πώ θα χρηματοδοτηθούν οι προτεραιότητε τη ενεργειακή στρατηγικής, Αυτό είναι αποφασιστική σημασία και λαμβάνοντα υπόψη το πακέτο Juncker και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και το καθεξής. Και τέλο το έκτο σημείο είναι γεωπολιτικού χαρακτήρα. Όπω είπε ο κ. Σαλντάργκα, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ένα εξόπιστο εταίρο η Ρωσία, αλλά και η εξάρτηση του κάθε κράτου δεν αφορά μόνο το αέριο. Η επενδύσει των Ρώσων στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα είναι πολύ μεγάλη, ακόμα και στον τομέα των πυρηνικών. Να μην το ξεχνάμε λοιπόν. Δεν μιλάμε μόνο για Ρωσία. Εάν σκεφτούμε ότι μπορεί να έχουμε και άλλους αναξιόπιστους εταίρους σε άλλες περιοχές του κόσμου, καταλαβαίνουμε ότι δεν ε, προωθούμε την ενεργειακή μας ασφάλεια, απλώς άλλου είδους εξαρτήσεις από άλλους αναξιόπιστους εταίρους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε συνάδελφε. Ο κύριος Ταμπουράνο από την EFTD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είχα καταλάβει ότι έχουμε τόσο χρόνο στη διάθεσή μα, γιατί θα είχα ετοιμάσει διεξοδικότερη παρέμβαση. Τέλος πάντων. Αυτό που με ευνηδίασε πάνω απ' όλα, διαβάζοντας αυτή την ανακοίνωση, είναι ότι το από το έγγραφο αυτό αποουσιάζει τελείως η διάσταση του πληθυσμού. Λέει πιο, ε, πιο πολλές υποδομές, οι άνθρωποι όμως ο κόσμο, όπω του ονομάζουμε εμεί στην Ιταλία, δεν αναφέρονται. Για να έχουμε μια πραγματική ενεργειακή ασφάλεια και αντεκτικότητα, οι διάφορε ομάδε του πληθυσμού θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι ενημερωμένε για του οικονομικού και πολιτικού κινδύνου που ε, όπου εκτιθέμεθα στην Ευρώπη λόγω της ενεργειακής μας εξάρτησης. Οπότε, πολύ περισσότερο από ότι στις υποδομές και στα τεχνικά στοιχεία θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις συνήθειες του κόσμου. Το κοινωνικό software, όπως θα τολμούσα να το πω. Και για το έγγραφο αυτό καθεαυτό, να πω ότι συμφωνώ με την ανάγκη μεγαλύτερης διασύνδεσης και διαφοροποίησης της προμήθειας, διότι αυτό πάντοτε τονώνει την ανθεκτικότητα, αλλά πρέπει να προσέξουμε και να μην οδεύσουμε προς μια υπερβολική ε, δυνατότητα στις υποδομές. Χρειάζονται πολλά στρατηγικά προγράμματα και θα πρέπει να δώσουμε έμβαση στις υποδομές, στις μεταφορές και την αποθήκευση των ρηκτών καυσίμων. Πρέπει να έχουμε περισσότερα προγράμματα για τα ευθύ δίκτυα και ως προτεραιότητα το να είναι αποτελεσματική χρήση των ε, κτηρίων του κατασκευαστικού τομέα στην Ευρώπη που πολλές φορές αυτή τη στιγμή ενεργειακά δεν είναι σωστά εξοπλισμένο, βασίζεται στο αέριο και οδηγεί σε περιπτώσεις ενεργειακής φτώχεια, ιδίω για τις μειονεκτούσες κοινωνικέ τάξεις. Ξέρουμε ότι το αέριο από το οποίο είμαστε εξαρτημένοι μαζικά και σε μεγάλο βαθμό, στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται για την θέρμανση των κτηρίων. Επίσης, η σταθερότητα είναι απαραίτητη για να έχουμε ανθεκτικότητα και αποδοτικότητα. Τη σταθερότητα όμως από ιστορικής πλευράς δεν μπορούμε να την εγγυηθούμε, διότι η προμήθεια ενέργειας έρχεται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές με πολύ σοβαρά γεωστρατηγικά προβλήματα, όχι μόνο τη Ρωσία και την Ουκρανία. Ε, ας θυμηθούμε τα διαδάγματα της ιστορίας. Επίσης, οι υποδομές της πετρελαιοβιομηχανίας πέραν του αερίου είναι πολύ σημαντικές. Δεν είναι εγγυημένη όμως η προμήθεια σε πετρέλαιο, διότι και το πετρέλαιο ε, πολλές φορές γνωρίζει διακυμάνσεις μη αναμενόμενος όπως η χαμηλή τιμή του ε, πετρελαίου αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει να στηρίξουμε την διεθνή παραγωγική δυνατότητα, κοιτάζοντας τα κοιτάσματα που έχουν ε, ανακαλυφθεί πρόσφατα, κοιτάζοντας πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τη σωστή αξιοποίησή τους μακροπρόθεσμα και χωρίς να υπάρχουν οι σημερινές ε, αναταράξεις της παγκόσμιας προμήθειας. Να μην ξεχνάμε άλλωστε και την κρίση που έχει προκύψει από το 2008 με, την, ε, με το σχιστολιθικό αέριο και αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε Shell Prime. Να κοιτάξουμε επίσης τις εγχώριες πηγές, ε, τις εγχώριες δυνατότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην Ευρώπη με τα ορυκτά δεν είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την δική μας κατανάλωση. Και μια τελευταία παρατηρήση, αν με επιτρέπετε πρόεδρε, δεν βλέπω καμία ασφάλεια να προκύπτει από το σύστημα ε, εξαρτησής μας από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Είδαμε πόσο ασταθές είναι εκεί το περιβάλλον, είδαμε τους πυρηνικούς σταθμούς που μπορεί να είναι ένας μόνιμος κίνδυνος για την Επιρώμα μας και θα έπρεπε να κλείσουν τελείως. Ευχαριστούμε κυρία Καστήγιο Βέρα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αναφέρθηκαν πάρα πολλές πτυχές του θέματος που μας καλύπτουν απολύτως. Ε, δεν πρέπει να μακρηγορήσω λοιπόν και εν συντομία θα προσπαθήσω να εστιάσω το ενδιαφέρον μου στη βάση του έργου αυτού κατά τη γνώμη μου. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Σαοντάργας γιατί η πρότασή του είναι πάρα πολύ περιεκτική. Ε, είναι πολύ σφαιρική η προσέγγιση του ε, στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Όλα αυτά που μας είπε βεβαίως πρέπει να περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε πρόταση για την ενεργειακή ασφάλεια και βεβαίως πρέπει να πω ότι εγγυόμαστε την ασφάλεια με τρεις τρόπους. Πρώτον, δεν έχουμε εξάρτηση, άρα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις ενεργειακές μας πηγές προμήθευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις με το να βρούμε νέες πηγές προμήθευσης και σε άλλες περιπτώσεις με το να έχουμε καινοτομία και τεχνολογία για να επιταχύνουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό καταρχάς. Δεύτερο, να υπάρχει σωστό σύστημα διασύνδεσης σε όλη την Ευρώπη. Και Ευχαριστώ τον κύριο Φόξ γιατί ανέπτυξε αυτό το θέμα που απασχολεί την Ισπανία. Και τέλος, να υπάρχει αποτελεσματικότητα στη λειτουργία όλων αυτών των συστημάτων διασύνδεσης, να λειτουργούν δηλαδή, να μην τα φτιάξουμε μόνο και μόνο για να υπάρχουν, αλλά όταν κληθούν να παίξουν το ρόλο τους να μπορέσουν να το παίξουν. Και γι' αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε το smart grid την έξυπνη σύνδεση σε δίκτυο. Θα πρέπει λοιπόν η ενέργεια να είναι ασφαλής, να είναι επαρκής δηλαδή, ασφάλεια με την έννοια της επάρκειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έρθει σε λίγο ο Επίτροπος Ενέργειας και αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και θα έχουμε τη δυνατότητα να του θέσουμε ερωτήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Πόσο μάλλον που έχουμε υπόψη μας το σχέδιο το επενδυτικό του Πρόεδρου Γιούνκερ ύψους 315 δις ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, ε, είναι μια πρώτη δυνατότητα να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μιγκελάρια Κανιέτε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να μιλήσουμε ε, για έργα που έχουν να κάνουν με υποδομές ενεργειακές και άλλες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ η κυρία Καρίμα, η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ. Να δηλώσω καταρχάς πως ενδιαφέρομαι για την έκθεση αυτή, γιατί είμαι αρμόδια από τους σοσιαλδημοκράτες και για τα θέματα της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική η ανταλλαγή απόψεων για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η έκθεση αυτή. Προκειμένου να μπούμε και στο μυαλό των συναδέλφων της ε, Επιτροπής ΙΤΡΕ και να πω ότι συμφωνώ γιατί πιστεύω ότι η ενεργειακή ασφάλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις είναι από τους πιο σημαντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία. Και αυτό σημαίνει αφενός ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, αξιόπιστη αναγωνιστική πρόσβαση στην παγκόσμια, στους παγκόσμιους πόρους. Αλλά, από την άλλη, θα πρέπει να συμμορφωθούμε με τις μακροπρόθεσμες ε, στοχοθετήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση του άνθρακα και για την παροχή ενέργειας σε προσιτές τιμές. Όλοι γνωρίζουμε ωστόσο ότι σήμερα η Ευρώπη είναι από τους πιο μεγάλους αγοραστές ενέργειας και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται συντονισμένη, ενωμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με τους μέσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της που πιστεύω ότι χρειάζονται κατεπηγόντως. Και υπάρχουν και δύο βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει να υπογραμμίσουμε. Καταρχάς ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα, ότι τα προγράμματα προτεραιότητας θα πρέπει να επιταχυνθούν προκειμένου να αποφευχθούν η ενεργειακή νήση και επίσης ε, για να επιτευχθεί ο στόχος του 10% σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά, τις ηλεκτρικές υποδομές μέχρι το 2020 και ότι επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαφοροποιήσει τους παρόχους, τους προμηθευτές της ε, και σε ό,τι αφορά τον ε, νότιο άγωγο αερίου και τέλος να εκφράσω την υποστήριξή μου για την δομή των οκτώ πυλώνων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέσσερις εξ αυτών θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η διαφεροποίηση της παροχής και της υποδομής, η ανάπτυξη τεχνολογιών ενέργειας, η δημιουργία μιας εύρυθμα λειτουργούσης αγοράς και βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από δική μου πλευρά, λοιπόν, από πλευρά της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ε, είμαι στη διάθεση των συναδέλφων της Επιτροπής Ήτρα, προκειμένου να είναι συντονισμένη η δράση μας. Μιλάμε για κάτι που χρειάζεται και που χρειάζεται κατεπηγόντως. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Ντάλη. Ο κύριο Κάριν, είναι επόμενος ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά ακούσαμε. Στη δεκαετία του 70, με το εμπάρκο του πετρελαίου και την πετρελαϊκή κρίση, έγιναν κάποιες ε, πολύ σημαντικές αλλαγές σε όλο τον κόσμο. Η Γαλλία εισήγαγε πρινική ενέργεια, οι ΙΠΑ ξεκίνησαν μακροπρόθεσμοι αναζήτηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας, μάλλον αφελής, σε ό,τι αφορά τη χρήση ορεικτών πόρων. Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη, αλλά και όχι μόνο στην Ευρώπη, λαμβάνει μια νέα διάσταση με τη, τα γεγονότα του τελευταίου έτους, με την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία σε ό,τι αφορά τη χρήση και την εκμετάλλευση της ενέργειας ως πολιτικό εργαλείο για την επιρροή στην Ευρώπη. Παρόμοια με τη δράση της Ανατολής ε, στη δεκαετία του 70, στην πετρελαϊκή κρίση. 53% της συνολικής κατανάλωσης, 66% του πετρελαίου εισαγάγεται το πιο πολύ από τη Ρωσία και το ίμιση εξ αυτού εισαγάγεται μέσω της Ουκρανίας. Άρα είναι προφανές ότι υπάρχει υπερβολική εξάρτηση από μία και μοναδική πηγή ενεργειακής προμήθειας. Ποιες είναι οι λύσεις λοιπόν. Έχουν ήδη αναφερθεί. Ήθελα μόνο και εγώ να αναφέρω το πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Ο κύριος Φόξ και άλλοι έθεσαν το πώς έχουν τα πράγματα. Αλλά χρειαζόμαστε λοιπόν μια ενιαία εύρυθμα λειτουργούσα αγορά σε ό,τι αφορά θέματα ενέργειας. Η προσφορά από τη μία πλευρά θα μπορούσε να μεταφερθεί σε άλλον προμηθευτή. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε τα προγράμματα διασυνδεσιμότητας, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Χρειαζόμαστε διαφοροποίηση των πηγών. Θα πρέπει να βρεθεί μία λύση. προκειμένου να υπάρχουν ε, άλλοι πάροχοι προμηθευτές αερίου, που δεν θα είναι η Ρωσία. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή τον κύριο Σάντορκα, για τις αρχικέ αυτές σκέψεις και ιδέες. Αυτό που χρειαζόμαστε όμω είναι μία μετατόπιση και μάλιστα κατεπηγόντως όπως αυτή μετά το εμπάργκο της δεκαετίας του 70. Γιατί εξαρτώμαστε υπερβολικά όχι από τη Μέση Ανατολή και το πετρέλαιο πλέον, αλλά από τη Ρωσία. Και η Ρωσία συμπεριφέρεται απρόβλεπτα. Αυτό είναι γεγονός. Όσο και να μην μας αρέσει, θα πρέπει να το λάβουμε ως δεδομένο και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και να είμαστε λιγότερο εξαρτημένοι από τους εκβιασμούς τους ενδεχόμενου του μέλλοντος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, Βιντάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ενεργειακή ασφάλεια ως προς την ε, ασφάλεια της ε, παροχής και της προμήθειας είναι κάτι που απασχολεί τις ευρωπαϊκές πολιτικές από τη δεκαετία του 70 με τις κρίσεις του πετρελαίου του 73 και 79 Εκεί είδαμε πόσο υπερβολική ήταν η εξάρτηση της Ευρώπης από το πετρέλαιο του ΟΠΕΚ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η σημερινή κατάσταση μας υποχρεώνει και είναι ένας από τους στόχους μας, ε, αναγνωρισμένος μάλιστα στις συνθήκες, να δράσουμε. Η κρίση της Ουκρανίας δεν θα πρέπει κατά την άποψή μου να είναι ο μόνος λόγος που θα μας κάνει να αναλάβουμε δράση ωστόσο για την ενεργειακή μας ασφάλεια και αυτάρκεια. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού για την Ενέργεια υπολογίζει ότι μεταξύ 2010-2035 η διεθνή ζήτηση για ενέργεια θα αυξηθεί κατά το 1 τρίτο. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν αναφέρει μια βασική πρόκληση για την ενεργειακή μας πολιτική και μάλιστα με τρόπο ευθύ δεν παραλείπει καμία από τις επιλογές που διαθέτουμε για να τονώσουμε και να βελτιώσουμε την ενεργειακή μας αυτάρκεια. Αντί όμως να βάλει όλα τα ε, αυγά στο ίδιο καλάθι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τελικά προτείνει μια η ιεράρχηση των ε, στόχων. Καλά κάνει και δίνει έμφαση η ανακοίνωση τη Επιτροπή στο ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, διότι μπορεί να είναι εγχώρια προέλευσή του και σωστά δεν ξεχνά και άλλε συμπληρωματικέ οδού, όπω το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το σχιστολιθικό αέριο, την αποθήκευση και διατήρηση άνθρακα. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ε, απαρνηθεί την, τον οποιανδήποτε μικρό πόρο μπορεί να διαθέτει γιατί ε, οι εξαγωγές ε, πόρων θα, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουν υπόψη και την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση. Ε, στον τομέα της ενέργειας λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε να συγκεντρώσουμε το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων και για την έρευνα. Έτσι ώστε να έχουμε το πιο ανταγωνιστικό αηφόρο σύστημα προμήθευσης ενέργειας. Και επομένως η ανακοίνωση αναγνωρίζει και καλώς ότι είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουμε σωστά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη και τον Ορίζοντα 2020. Τέλος, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε την ενοποίηση ή την ολοκλήρωση του, της ενιαίας αγοράς ενέργειας. Είναι στόχος που είχε τεθεί για φέτος, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Είναι επίγον η διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών κατά 10%. Αυτό έχει επαναλάβει πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν θα πρέπει να είναι πια προγραμματική δήλωση. Πρέπει να περάσουμε στην πράξη. Αυτό απαιτεί το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου για το πλαίσιο για το 2020. Είναι δεσμευτικός στόχος. Και για να γίνει πραγματικότητα πρέπει να επενδύσουμε τα σύνορα, στις υποδομές, τις διασυνοριακές που συνδέουν τα νησιά με την κεντρική Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και να φτάσουμε στο 15% μέχρι το 2030. Και καλώς το τονίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι επειδή είμαι Ισπανός, αλλά επειδή είμαι Ευρωπαίος θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε στην Ισπανία πλεόνασμα στις δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έχουμε τους περισσότερους και μεγαλύτερους ε, τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου στους οποίους έρχεται φυσικό αέριο από διάφορες άλλες χώρες και μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που εξαρτώνται από φυσικό αέριο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο Herbert Ρόιλ, παρακαλώ, έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, Εδώ και αρκετό καιρό μιλάμε για την ενέργεια στην Ευρώπη και για το πόσο σημαντική είναι, αλλά σπάνια μιλάμε για την ε, ασφάλεια εφοδιασμού. Η ασφάλεια εφοδιασμού λοιπόν είναι πολύ βασική. Τα τελευταία χρόνια ασχοληθήκαμε με πολλές άλλες πτυχές της ενέργειας για τις επιπτώσεις ε, στο κλίμα και το καθεξής, αλλά έχουμε παραμελήσει αυτή την διάσταση και πλέον ε, τα πράγματα ζορίζουν. Θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις οι απαντήσει άλλωστε δεν είναι τόσο περίπλοκες, αν ε, συνοψίσουμε αυτά που ακούσαμε σήμερα. Ποτέ δεν μπορούμε να βγάλουμε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Το είπε και ένα συνάδελφο, ε, ούτε ένα πάροχο, ούτε ένα είδο μονέργειας μόνο, προκειμένου να υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις σε περίπτωση ανάγκης. Και γι' αυτό λοιπόν η είναι ανοησία ασφαλώ να πιστεύουμε και είναι και επικίνδυνο να πιστεύουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον μόνο ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Θα πρέπει να συζητάμε και άλλε ε, και τα άλλα μέσα. Ή τουλάχιστον όσο υπάρχουν να μην τα αφήνουμε κατά μέρο. Οι Αμερικανοί μα δείχνουν πώ μπορούν να εξορίσουμε πετρέλαιο με πιο μοντέρνου τρόπου. Στην Ευρώπη απλά δεν τα λαμβάνουμε υπόψη αυτό. Και μένουν να χρησιμοποιείται οι πόροι που βρίσκονται στη γη στην Ευρώπη και δεν ξεκινάει η συζήτηση για το φρέκινγκ για παράδειγμα, για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το για τη μέθοδο της υδρορογμάτωσης για την εξόρυξη. Πολύ λυπάμαι, αλλά όποιος θέλει ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και ασφάλεια εφοδιασμού και μια ισχυρή βιομηχανία αλλά και για τους πολίτες. Αν θέλουμε λοιπόν την ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει να έχουμε ευρύ, ευρία γκάμα για τη χρήση των μελλοντικών ε, τεχνολογιών αλλά και των παραδοσιακών τεχνολογιών. Αυτό αν γίνει μετά από πολιτικές διαβουλεύσεις το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα καλό. Αν περιοριστούμε μόνο στι ε, στις πηγέ πηγές ενέργειας θα έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ συνάδελφε. Επόμενο και τελευταίος ομιλητής στη λίστα, ο συνάδελφος Μαρινόφ. Ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο, διότι υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις. Είναι πραγματικά πολύ αρνητικό που ακυρώθηκε το πρόγραμμα του Νότιου Διαδρόμου. Ως βούλγαρος εκπρόσωπος εδώ ε, εγώ πρέπει να πω ότι δεν συμφωνώ καθόλου με την απογοήτευση που εκφράστηκε. Για τρία χρόνια ε, οι ρωσικές αρχές πίεζαν την Βουλγαρία να παραβιάσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για να ξεκινήσει την οικοδόμηση αυτού του αγωγού. Ευτυχώς ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε τρεις βουλγαρικές κυβερνήσεις η μία μετά την άλλη δεν ακολούθησαν αυτές τις πιέσεις, δεν υπέκυψαν. Ε, καταφέραμε ο κύριος Πούτιν να παραδεχθεί ότι ένα κράτος δικαίου υπάρχει, ότι υπάρχει ένα νέο ενεργικό πακέτο και ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Βεβαίως τώρα θα υπάρξουν πιέσεις πάλι στη βουλγαρική κυβέρνηση και τους βουλγαρούς πολίτες, διότι με το παραμικρό πρόβλημα στην ενέργεια τα το σφάλμα θα επιρριφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν επιτρέπει να παραβιαστούν οι νόμοι της. Δηλαδή είναι πολύ υψηλό το διακύβευμα. Αυτό που θα επιχειρήσει τώρα η Ρωσία την ερχόμενη τριετία είναι τελείως προβλέψιμο. Θα φροντίσει να ε, μειώσει το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξηγώντα τους πολίτες ευρωπαϊκών χωρών ότι ό,τι πρόβλημα έχουν φταίει γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι έχουμε αυστηρούς κανόνες που δεν θέλουμε να τους ε, παραβούμε, να τους κάνουμε πιο ευέλικτους για να συνεργαστούμε μαζί τους. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε εναλλακτικέ και λύσεις που θα πρέπει να προταθούν σε λύσεις που τόσο πολύ εξαρτώνται από την ε, προσφορά των ε, Ρώσων. Οι αριθμοί ήδη αναφέρθηκαν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε συνάδελφε για τις παρατηρήσεις σας. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Χάνς Φανστέν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και όλα τα μέλη που έλαβαν το λόγο για, για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι μπορώ να είμαι σχετικά σύντομος. Αυτά που άκουσα ως τώρα ε, έχουν πολύ καλή θέση στην έκθεση. Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της άλλωστε. Και Ελπίζω να έχω συνομιλήσει με τον κύριο Σοντάργα σύντομα. Όμω, τα βασικά στοιχεία τη ε, στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον ένα τον άλλο τρόπο έχουν αναφερθεί στη σημερινή απογευματινή συζήτηση. Η δυσκολία είναι να τα ανακεφαλαιώσει κανεί, να τα συμπεριλάβει στην έκθεση με τρόπο που να είναι ισόρροπο, αλλά αυτό φαντάζομαι θα είναι αποτέλεσμα του κοινού έργου των μελών αυτή τη Επιτροπή. Ένα σημείο θα ήθελα να σχολιάσω ένα σημείο στο οποίο δεν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις σημερινές συζητήσει. Η ευρωπαϊκή διάσταση της ενεργειακής ασφάλειας από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθήσαμε το μήνυμα αυτό να ε, περάσει ξεκάθαρα από τη στρατηγική. Και αυτό επιβεβαιώθηκε και από το έργο που κάναμε με τα τεστ κόπωσης για το αέριο η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης είναι πραγματικά ένα ζήτημα ευρωπαϊκό και θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ε, εξετάζεται. Τα κράτη-μέλη προσπαθούν να ε, λύσουν τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας μονομενα, αλλά εάν κάνουν κάτι τέτοιο και πιο ακριβά θα πληρώσουν και λιγότερο αποτελεσματικό θα είναι ε, θα και πιο λιγότερο αποτελεσματική θα είναι προσπάθεια και δεν θα έχουν φτηνή και εύκολα προσβάσιμη ενέργεια για τους πολίτες. Υπό αυτή λοιπόν την πρόπτικη θα πρέπει να περάσει αυτό ισχυρό μήνυμα μέσα από την έκθεση και από το Κοινοβούλιο ε, ενώ και θα πήγαινα και πιο μακριά λέγοντα ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα τη Ευρώπη των 28 ή των 100 μελών. Πρέπει να το δούμε από την ευρύτερη πρόπτικη που θα συμπεριλαμβάνει την ενεργειακή κοινότητα συνολικά και τι χώρε γειτονία τη Ευρώπη. Διότι και αυτά είναι στοιχεία που καθορίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της Επίρου. Ξέρω ότι θα έρθει σε πολύ λίγη ώρα ο Επίτροπος Κανιέται, οπότε θα παραμείνω σε αυτά τα σχόλια για την ώρα. Και απλώς να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε αποσαφήνιση μπορεί να χρειαστείτε. Για οποιαδήποτε πτυχή της έκθεσης. Θα αναμένουμε τη συνέχεια της συζήτησης στο Κοινοβούλιο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Εκπρόσωπε της Επιτροπής. Ας πάμε στον ε, αρμόδιο εισηγητή μας, τον συνάδελφο Αλγκύρντας Σαουντάργας, για την τελική σας παρέμβαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση αυτή. Όπως ε, προανέφερα, μετά την ανταλλαγή απόψεων με τους κοιόδης εισηγητές θα προσπαθήσουμε και ήδη σε έναν βαθμό θα ενσωματώσου, έχουμε ενσωματώσει ιδέες στο σχέδιο έκθεσης καλύπτοντας όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν. Θέλουμε να δούμε το θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες αλλά να κάνουμε και αυτό που πολύ σωστά εντόπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή να έχουμε ένα ισόρροπο αποτέλεσμα. Καλύπτοντας όλα τα ζητήματα ουσίας. Αυτά που αναφέρθηκαν εδώ, σχεδόν όλα, ούτως ή άλλως, με τον ένα τον άλλο τρόπο είναι πολύ σημαντικά ή αν τα δει κανεί από διαφορετικέ κοπιές. Γι' αυτό έχω παραμείνει σε λίγε παρατηρήσει, κάπω πιο γενικέ, αλλά για συγκεκριμένα ζητήματα. Λόγω χάρη, όπως αναφέρθηκε, η ενέργεια είναι σημαντική και για τη βιομηχανία, αλλά και για του πολίτε. Είναι σαφέ αυτό. Και αυτή, αυτός είναι και ο ορισμός της ε, ενεργειακής ασφάλειας στην ουσία του κοινωνική συνιστόσα θα περιλαμβάνεται στην έκθεση και ε, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις για την καταπολέμηση της ενεργειακής ε, φτώχειας αλλά δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα μία μόνο έκθεση. Να προτείνει δηλαδή λύσεις για όλα τα προβλήματα. Αυτή και μόνο η έκθεση. Παρόλο που το κοινωνικό σκέλος το ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι. Ίσως δεν το τόνισα αρκετά στην αρχική μου παρουσίαση, η αγορά είναι ο βασικός τρόπος για να ε, διασφαλίσουμε το μέλλον. Όμως το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά, αν όχι καθημερινά, πάντως πολύ στενά για το θέμα αυτό. Θα συνεχιστεί λοιπόν η όλη συζήτηση και να μην συμφωνήσω με τον συνάδελφο Γιάβορα απλώς, λέγοντας ότι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 ότι όλα αυτά ίσως να μην έχουν ε, μεγάλη σημασία πια γιατί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προταθεί και τελείωσε. Δεν συμφωνώ. Τα συζητήσαμε και στην συνάντησή μας και θα τα επαναλάβω και εδώ. Νομίζω ότι ο διάλογος αυτός είναι διάλογος διαρκείας μέχρι να εγκριθεί ε, και να συμπεριληφθεί η Ευρωπαϊκή Στατική Ενέργεια στην νομοθεσία της Ένωσης ως ένας πυλώνας της, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε ακόμη. Και, και άλλες πτυχές αναφέρθηκαν, όπως αυτό που έγινε πρόσφατα με τον νότιο διάδρομο. Δεν αναφέρεται πλέον ο νότιος διάδρομος, το South Stream στην έκθεσή μας. Ούτε ο Ναμπούκο. Άλλα α, ε, προγράμματα θα πρέπει να αναφερθούν. Όχι το South Stream όμως, ούτε το Ναμπούκο. Φοβούμαι ότι η Ρωσία έχει όντως κάποια, κάποιες στην περιοχή. Ακούσαμε και τι έγινε με την Τουρκία. Ο Πούτιν δεν σκέφτεται μόνο τον Blue Stream που ήδη λειτουργεί, αλλά τελικά σκέφτεται και το South Stream να επηρεάσει για να περάσει από την ε, Μικρασία. Εάν δεν είμαστε λοιπόν αποφασιστικοί και δεν δείξουμε πυγμή, ό,τι έγινε ε, στην ε, περίπτωση του Ναμπούκο θα γίνει και στην ε, μικρά ουσία και θα έχουμε ένα Πουτινούκο, για να σας το πω και λιθουανικά, ένα μικρό Πούτιν δηλαδή. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Το ανέφερε η κυρία Καστιλιαβέρα τα έγγραφα. Να σας πω ότι όλα είναι διαφανή γιατί ο συνάδελφος εισηγητής μοίρασε μία σελίδα σε όλους τους κοιοδείς. Όλα λοιπόν είναι απόλυτα διαφανή. Δεν είναι ακόμα το σχέδιο έτοιμο, το σχέδιο έκθεσης. Θα ετοιμαστεί σε κάποιες ημέρες, σε κάποιες εβδομάδες, ίσως πριν τα Χριστούγεννα, πώς σας εξαρτάται το σχέδιο της έκθεσης ε, το οποίο και θα εξετάσουμε στις 21 Ιανουαρίου του 2015 προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Επτά ημέρες αργότερα 28 Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι. Εξέταση των τροπολογιών στις 23 Φεβρουαρίου του 2015, στις 14 Απριλίου ψηφοφορία στην Ήτρε, στην Ολομέλεια ΔΕ το Μάιο του 2015. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα για την έκθεσή μας για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια. Τώρα χρειαζόμαστε να κάνουμε διάλειμμα τριών λεπτών γιατί έχει καταφτάσει ο Επίτροπος και θα χρειαστεί τρία λεπτά μέχρι να έρθει στην αίθουσα. Ευχαριστώ. Τρία λεπτά διάλειμμα.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 Yeah. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Φίλοι μου, κυρίες και κύριοι. Δεν αρχίζει τώρα η χριστουγεννιάτικη δεξίωση. Θέλουμε ακόμα να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Έχουμε να συζητήσουμε. Δεν ξέρω και τι να κάνω. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, μετά την ε, ταραχώδη ακρόαση στην Επιτροπή μας, περνάμε τώρα στο διαστρωμένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαστρωμένος διάλογος. Πρώτος τη τάξη, ο Επίτροπος για το κλίμα και την ενέργεια. Καλά τα είπα με αυτή τη σειρά. Όχι κλίμα και ενέργεια, ενέργεια και κλίμα. Με συγχωρείτε, αλλάζω λίγο τον τίτλο του χαρτοφυλακίου σας, κύριε Επίτροπε. Να πω τα εξής. Τι είναι το σημαντικό για μας. Η σημερινή ανταλλαγή απόψεων είναι μέρος του λεγόμενου διερθρωμένου διαλόγου με την διθεσμική συμφωνία Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Βασικός σκοπός είναι να συζητηθούν οι προτεραιότητες της πολιτικής ενέργειας και η συμπερίληψη στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως θα πρέπει να μην ξεχνάμε και τα θέματα του κλίματος και τα σχετικά μέτρα, διότι είμαστε υπεύθυνοι για το συνδυασμό των μέτρων για την ενέργεια και αυτών για το κλίμα. Κυρίως διότι η διάσκεψη των μερών υπαριθμών 20 στη Λίμα ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες, τρεις μέρες για την ακρίβεια. Κάποιοι από εμά θα πάμε στη Λίμα την ερχόμενη εβδομάδα και εγώ ίδιος. Οπότε δεν θα είμαστε όλοι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλα μπορεί να ανακύψουν. Γιατί έχουμε τον ε, Επίτροπο που είναι υπεύθυνο και για τα δύο θέματα, και το κλίμα και την ενέργεια. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία μα, στην ιστορία του Ευρωκοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, που αυτά τα θέματα συνδυάζονται. Ίσως έτσι να είναι πιο ε, επικοδομητική η προσέγγιση από όλες τις πρόπτικες. Παρακαλώ λοιπόν τον κύριο Μιγγέλα Κανιέτε να λάβει το λόγο για την ομιλία του. Προκαταρκτική, εισαγωγική μάλλον ομιλία για όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Γέρση. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Στην Επιτροπή μιλάω αγγλικά αλλά σε αυτή την περίπτωση θα μιλήσω ισπανικά. Καλησπέρα σε όλους. Για μένα είναι μεγάλη χαρά να παίρνω το λόγο εδώ για πρώτη φορά στην Επιτροπή σας με την ιδιότητά μου ε, του Επιτρόπου για την ενέργεια και την δράση για το κλίμα. Όπως γνωρίζετε, στην Ακρόαση, όταν ήμουν υποψήφιος Επίτροπος, δεσμεύτηκα να ξεκινήσω έναν πολύ ε, ειλικρινή και έντονο διάλογο με εσάς και γι' αυτό θέλησα να έρθω ε, ενώπιόν σας για να σας μιλήσω για το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα, αξιότιμοι βουλευτές, φαίνεται περισσότερο από κάθε φορά το γεγονός ότι η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται άρρηκτα με την ευημερία των πολιτών και της, του συνόλου της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Και γι' αυτό το λόγο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θεωρεί ότι μία ενεργειακή ένωση Ένωση με πολιτική σωστή για την ε, κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα παραδοτέα που θα πρέπει να μπορεί να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γι' αυτό η παρουσίαση για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα παρουσιάσουμε στις αρχές της επόμενης χρονιάς θα είναι φιλόδοξη και θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή σε αυτό το τομέα. Περισσότερη Ευρώπη σε αυτό το κλάδο είναι η πολύ σημαντική πρόκληση που υψώνεται μπροστά μας. Το έργο για την Ενεργειακή Ένωση το συντονίζει ο Αντιπρόεδρος Σεύκοβιτς και βασικός στόχος είναι να πετύχει καταρχάς την ανταγωνιστικότητα την οποία επιθυμούν, την οποία έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις μας. Και έτσι οι ενεργειακές τιμές, οι τιμές της ενέργειας πρέπει να είναι προσβάσιμες και για τα νοικοκυριά και για τη βιομηχανία και να είναι συγκρίσιμες με αυτές των ανταγωνιστών μας. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε διαφοροποίηση εσωτερική και εξωτερική διαδρομών προμήθευσης πηγών ενέργειας και ε, και διαφόρων προμηθευτών ούτως ή άλλως. Ε, αυτό είναι απαραίτητο για να έχουμε καλύτερη πορεία και να μπορέσουμε να έχουμε αλληλεγγύη με τις επόμενες γενιές. Η Ενεργειακή Ένωση, είπε ο Αντιπρόεδρος Σεύκοβιτς, θα εδράζεται σε πέντε βασικούς πυλώνας. Πρώτον, η επάρκεια της προμήθευσης με βάση την αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη. Δεύτερον, η ανταγωνιστικότητα και η αποκορύφωση, αν θέλετε, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Τρίτον, ο εξυγχρονισμός της ζήτησης και η ενεργειακή εξοικονόμηση. Και τέλος, θα πρέπει να μιλήσουμε για την έρευνα αλλά και για την ανάπτυξη. Θα ήθελα όμως να προσθέσω εδώ ένα πολύ σημαντικό πυλώνα, την εσωτερική αγορά ενέργειας. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ανοιχτή και ανταγωνιστική, με κανόνες οι οποίοι να εφαρμόζονται και να υπάρχει φυσική διασύνδεση, ηλική διασύνδεση δηλαδή όχι μόνο επί χάρτου και θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια για να υπάρξει πραγματική εσωτερική ενιαία αγορά ενέργεια. Από πλευράς κανονιστικών διατάξεων έχουμε σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει να εγγυηθούμε τώρα τη σωστή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, των υφιστάμενων κανόνων, γιατί μόνο έτσι θα είμαστε σε θέση να υποβάλουμε νέες προτάσεις με έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει ότι το τρίτο ενεργειακό πακέτο θα πρέπει να είναι πλήρως καταρτισμένο στα τέλη του 2014 και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι σε αυτό το σημείο. Θα κάνω το παν, δεν θα διστάσω εάν κληθώ να επιβεβαιώσω ότι όλα τα κράτη ε, έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους ως προς την ενσωμάτωση στο ε, εθνικό δίκαιο του κοινοτικού δικαίου. Είτε πρόκειται για μεγάλα κράτη, είτε πρόκειται για μικρά κράτη και για το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και για ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Θα ε, βεβαιωθώ ότι όλοι συμμορφούνται και όλοι προχωρούν με τη σωστή ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής νομοθεσίας. Όλα αυτά θα είναι σημαντικά γιατί έτσι θα έχουμε καλύτερη τεχνική βοήθεια όταν έχουν αμφιβολίες τα κράτη-μέλη για το πώς θα εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και έτσι θα μπορέσουμε να σιγουρευτούμε ότι όλοι συμμορφούνται με τους ίδιους κανόνες. Πέραν όμως της κείμενης νομοθεσίας πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν οι απαραίτητες διασυνδέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ενιαία εσωτερική αγορά ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει αρκετά, επιλέγοντας έργα κοινού ενδιαφέροντος, κοινού συμφέροντος. Έχουμε εντοπίσει 248 έργα κοινού ενδιαφέροντος και 72 από αυτά έχουν οριμάσει αρκετά, μπορούν να οριστικοποιηθούν το 2017. Υπ' αυτή την έννοια το σχέδιο Juncker που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα είναι ένα πολύ καλό νέο. Ενισχύει το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια ευκαιρία για να έχουμε καλύτερες ενεργειακές υποδομές, για να μειωθεί το κόστος και είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι αρκετά ευέλικτο. Μπορεί να περιλάβει νέα έργα κοινού ενδιαφέροντος έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο του 10% της ηλεκτρικής διασύνδεσης του 2020, το 15% το 2030 και να έχουμε μεγαλύτερη διαφοροποίηση εξωτερικών προμηθευτών ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο φυσικό αέριο. αέριο. Θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωση σχετική για το πώς θα πετύχουμε αυτό το στόχο της διασύνδεσης του 10% και του 15% αντιστοίχως σε βάθος χρόνου. Επιστρέφω όμως στο επενδυτικό σχέδιο του Προέδρου Γιούγκερ και θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν είναι μόνο ένα μέσο επενδύσεων σε υποδομές. Λαμβάνει υπόψη και την κινητοποίηση πόρων στον τομέα και στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Λαμβάνει υπόψη την ενεργειακή αποδοτικότητα, την έρευνα και την καινοτομία. Και αυτοί είναι οι θεμελιώδεις πυλώνες που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε το στόχο μας, το στόχο μας που είναι η μείωση των εκπομπών αερίου που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μεταξύ άλλων θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Το κλίμα ε, είναι η μία πλευρά του νομίσματος και η ενέργεια είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Αν έχουμε ένα αηφόρο ενεργειακό σύστημα, τότε θα έχουμε πολύ καλή πρόοδο και σε οικονομικό επίπεδο και στον αγώνα για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Η Ενεργειακή Ένωση είναι ευκαιρία για να, μια, να δώσουμε μια νέα οικονομική και πολιτική όθηση στην Ευρώπη. Επομένως, το πλαίσιο δράση σε θέματα κλίματος και ενέργειας μέχρι το 2030, ένα πλαίσιο που αποφασίστηκε στο περασμένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι στόχοι είναι πολύ γνωστοί σε εσάς. Μιλούμε για 40% μείωση των εκπομπών, 27% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 27% ενεργειακή αποδοτικότητα καλούμεθα και υποχρεούμεθα να έχουμε πιο συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γι' αυτό θα έχουμε ένα σύστημα διακυβέρνησης το οποίο θα στηρίζεται πρώτο στα εθνικά σχέδια των κρατών μελών και δεύτερον στις ευρωπαϊκές δράσεις. Και το ένα και το άλλο. Το σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης πρέπει να είναι αξιόπιστο, πρέπει να είναι διαφανές, να δίνει ευελιξία στα κράτη-μέλη, να έχουν αυτά την ελευθερία να αποφασίσουν το ενεργειακό τους μείγμα. Πρέπει να προβληματιστούμε πώς θα υλοποιήσουμε αυτή τη σωστή διακυβέρνηση, πώς θα υπάρχει συνοχή αρχή στο σχεδιασμό και πώς θα ελέγξουμε και θα επαληθεύουμε και θα αξιολογούμε την πρόοδο του καθενός. Θέλουμε, θέλω να προχωρήσω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και σκοπεύω να παρουσιάσω συγκεκριμένη πρόταση το πρώτο εξάμεινο του 2015. Η Ενεργειακή Ένωση πρέπει να είναι μέσο για να αναζωπηρωθεί η οικονομία. Πρέπει αυτό το πλαίσιο και αυτός ο στόχος να το θεωρήσουμε ευκαιρία για τη βιομηχανία μας. Να το πω αλλιώς, πρέπει να είναι ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη εάν λειτουργήσουμε και δράσουμε έξυπνα. Υπ' αυτή την έννοια, το σύστημα εμπορίας αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και εκπομπών σχετικών ε, σχετίζεται άμεσα με τη βιομηχανική ε, αηφορία και είναι ακρογωνίως λίθος του συστήματος. Η βιομηχανία μας πρέπει να έχει τους απαραίτητους μηχανισμούς για να μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχουμε θέσει με ορίζοντα το 2030 και πέρα από αυτό. Ο σε αυτή την Επιτροπή ε, εγνωμοδότησε συντάσσει ο φίλος μου κύριος Αντώνιο Ταγιάννη, πρώην και είναι πολύ σημαντικό το κείμενό του. Ε, δίδεται σημασία στη σταθεροποίηση του συστήματος για την εμπορία ε, των εκπομπών των ρήπων θα ήθελα όλα αυτά να υιοθετηθούν το συντομότερο δυνατόν, γιατί μόλις εγκρεθούν θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε εμείς τη μεταρρύθμιση του συστήματος ε, εμπορίας εκπομπών και ρήπων και ιδανικά πριν το καλοκαίρι να γίνει αυτό. Αυτή η πρόταση πρέπει να εγκριθεί και θα ρυθμίσουμε το καθεστώς κατανομής δωρεάν δικαιωμάτων στη βιομηχανία αναλόγως με τις προσταγές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα λάβουμε υπόψη σε πολύ μεγάλο βαθμό βαθμό τις ιδέες της δικής σας κοινοβουλευτικής επιτροπής και θα τις έχουμε πάντοτε υπόψη μας και θα έχουμε πολύ σημαντικές επαφές μαζί σας πριν διατυπώσουμε τη νέα μας πρόταση. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την αναζωπήρωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ως προς τα νομοθετήματα για τους κλάδους που δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και ρήπων, ε, θα κάνουμε μια πολύ λεπτομερή αξιολόγηση καθ' όλη τη διάρκεια του 2015. Στην αξιολόγησή μας θα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία στα οποία μας έχει εφιστήσει την προσοχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου. Θα έχουμε ε, ιδιαίτερη μέρη γιατί για τον τομέα της γεωργίας, της χρήσης της γης, Επομένως, οι κλάδοι που δεν μπαίνουν στο σύστημα εκπομπής ρήπο ε, δεν θα μπουν στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέτος, αλλά βεβαίως έχουν τις ίδιες πιθανότητες και περισσότερες ακόμα να μπουν στο πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για τα επόμενα χρόνια. Θα υπάρξει μια διάσκεψη υψηλού επίπεδου πριν το καλοκαίρι για να υπάρξει περισσότερος προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο ο κλάδος αυτός μπορεί να συμβάλλει στο συλλογικό μας στόχο που είναι ε, η μείωση των εκπομπών. Ε, αερίων. Αναφέρομαι στη διάσκεψη με την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία είναι ένας κλάδος ο οποίος μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και οφείλουμε να έχουμε διάλογο, να φτάσουμε σε συνένεση με τον ευρύ κλάδο με της αυτοκινητοβιομηχανίας για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και γι' αυτό θέλουμε διάσκεψη υψηλού επίπεδου με ισχυρή εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ισχυρή παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις παγκόσμιες εξελίξεις έχουμε νέους στόχους για τις εκπομπές, τους έχουμε εγκρίνει και έτσι οι ανταγωνιστές μας λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο. Πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συνέχεια. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία και τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια που εισάγουμε. Περισσότερο από τα μισά από αυτά που καταναλώνουμε από πλευράς ενέργειας είναι ενέργεια εισαγόμενη. Επομένως, ε, είναι αυτό μια ευκαιρία και για την ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το να λύσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να έχουμε διαφοροποίηση προμηθευτών, πρέπει να διαφοροποιήσουμε και την κατανάλωσή μας και να αρχίσουμε να καταναλώνουμε με καλύτερο τρόπο. Η ενεργειακή επάρκεια λοιπόν θα είναι πυλώνας της πολιτικής μας για κάθε 1% εξοικονόμηση σε ενέργεια που επιτυγχάνουμε, εξοικονομούμε 2 ή 3% σε εισαγωγές φυσικού αερίου από σήμερα μέχρι το 2030. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορούμε να μειώσουμε κατά 22% ε, τις εισαγωγές σε φυσικό αέριο το 2030 εάν ε, πετύχουμε ε, αυτή την εξοικονόμηση σε σχέση με τα νούμερα και τα στοιχεία του 2010. Αν αρχίσουμε δηλαδή και να καταναλώνουμε πιο έξυπνα και να διαφοροποιούμε τις πηγές προμήθευσης. Έχουμε ε, το τρίτο σχέδιο τριετών εργασιών. Ε, θα το παρουσιάσουμε. Θα παρουσιάσουμε επίσης ε, αναθεώρηση αυτού στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Είναι αυτές οδηγίες που επιτρέπουν στα ε, ε, νοικοκυριά να έχουν εξοικονόμηση στην κατανάλωση της τάξης των 110 δις ετησίως πρέπει να ενισχύσουμε την επικοινωνία έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι, να μην θεω... Ευρωπαίοι πολίτες να μην θεωρήσουν ότι αυτό είναι παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ότι είναι μια συλλογική προσπάθεια για να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής, η ποιότητα ζωής. Καλό τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο να επικοινωνήσουν καλύτερα αυτή μας τη δράση. Η περασμένη... Στην περασμένη προεκλογική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ορισμένοι γελιοποίησαν αν θέλετε ε, τον αντίκτυπο της οδηγίας για το co-design. Όμως είναι το πιο σημαντικό εργαλείο που έχουμε για την ενεργειακή εξοικονόμηση. Σίγουρα μπορεί να έχουν διαπραχθεί και σφάλματα και λάθη. Όμως ο κατάλογος των προϊόντων που ενσωματώθηκαν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής είναι πολύ σημαντικός. Η οδηγία συμβάλλει στην ενεργειακή αποδοτικότητα, μειώνει τα τιμολόγια ενέργειας που πληρώνουν τα νοικοκυριά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να τη διατηρήσουμε την οδηγία αυτή και να την τελειοποιήσουμε, να την διορθώσουμε βεβαίω. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ε, ηγέτης στον τομέα αυτό και θα έλεγα ότι έχουμε επάρκεια ε, στην ε, προμήθεια ενέργειας από τη στιγμή που έχουμε ξυπνότερη και καλύτερη χρήση της ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, είναι πολύ σημαντικές. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να ενσωματωθούν καλύτερα στο σύστημα. Πρέπει να κάνουμε επενδύσεις σε έξυπνα δίκτυα, σε διασυνδέσεις, σε ε, τεχνολογίες αποθήκευσης της ενέργειας. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά και χρειαζόμαστε όλες τις πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μας σύστημα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ευκαιρία και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει το σωστό πλαίσιο για να αναπτυχθούν σωστά και θα υποβάλουμε πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Ορίστε κυρίες και κύριοι βουλευτές κάποιες από τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι στοιχείο κλειδί για την ενεργειακή επάρκεια, για την ενεργειακή ασφάλεια, ε, το οποίο, κάτι το οποίο είναι σημαντικό και κάτι το οποίο για να επιτευχθεί χρειάζεται περισσότερο συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το πακέτο το χειμερινό, το package ε, μας χρησιμεύσε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με την Ουκρανία φέτος το χειμώνα και αποκαθίσταται η απαραίτητη εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών για να μην βγει κανείς μας χαμένος. Πρέπει όλοι να συνεχίσουν να καταβάλουν προσπάθειες, να επιδεικνύουν ε, καλή διάθεση για να τα καταφέρουν όλα αυτά. Η εξωτερική διάσταση της ενεργειακής μας πολιτικής θα είναι ε, σημαντικό κομμάτι ε, των δράσεών μας. Κάνουμε προσπάθειες διαφοροποίησης όπως γνωρίζετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε τους εξωτερικούς μας προμηθευτές κατά τρόπο ώστε να ωφεληθούν όλοι οι Ευρωπαίοι. Ξέρω ότι πρόσφατα είχατε μία συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια και την ενεργειακή και επάρκεια. Και η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του κυρίου Σαουντάργας θα είναι ε, μια πολύ σημαντική ε, κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι καλό να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με περισσότερες λεπτομέρειες στο μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, ε, κλείνοντας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ την ανακοίνωση των ρωσικών αρχών βάσει της οποίας ακυρώνεται ο αγωγός South Stream. Σημειώνουμε την ε, απόφαση αυτή, την καταγράφουμε και θα αναλύσουμε την κατάσταση λεπτομερώς. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να σταθεροποιήσουμε την επάρκεια ε, προμήθευση στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη έτσι ώστε να επιτεχύνουμε την ένταξη όλων αυτών ε, των περιοχών στο, στα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε πολύ για τον νότιο αγωγό, το Southern Corridor και να προχωρήσουμε γρήγορα θα δουλέψουμε σκληρά τα επόμενα χρόνια και βασιζόμαστε στη δική σας στήριξη για να έχουμε επιτυχία στην αποστολή μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Αρμόδιε για το κλίμα και την ενέργεια. Και τώρα θα περάσουμε στους συντονιστές και άλλους συναδέλφους εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Κάριν για το ΕΛΚ. Ευχαριστούμε, κύριε Κανιέτε. Μέχρι εκεί φτάνουν τα σπανικά μου. Μπορώ να πω και μπαίνω δία. Και λίγες ακόμα λέξεις. Καλά. Λοιπόν, ας συνεχίσω στα αγγλικά. Ξέρω ότι τα καταλαβαίνετε. Πολύ ενδιαφέρουσα ατζέντα, πολύ ε, εντυπωσιακό το θεματολόγιο. Όμως προτού έρθετε, συζητήσαμε ακριβώς την έκθεση του κυρίου Σαουντάργκας για την ε, ασφάλεια της προμήθειας. Και συνδυαστικά με τους στόχους για το διοξίδιο του άνθρακα που αφορά πάλι το πρωτοφυλάκιό σας. Έχουμε πολύ διαφορετικές καταστάσεις αν μεταξύ των κρατών μελών στη χώρα μου την ε, Λετωνία είμαστε περίπου στο 3% των ανανεώσιμων, περίπου όπως η Σουηδία. Είμαστε πολύ ε, φιλικοί προς αυτά και κατά το 66% εξαρτημένοι από τη ρωσική ενέργεια. Ως προς την προμήθεια είμαστε εξαρτημένοι πολύ από τη Ρωσία. 100% του αερίου μας έρχεται από τη Ρωσία και είναι το 1 τρίτο της συνολικής μας κατανάλωσης στο αέριο. Το κράτος μέλος μας λοιπόν είναι τελείως, ε, σε τελείως παράδοξη κατάσταση. Τελείως πράσινο και τελείως εξαρτημένο. Ανασφαλές και μη αυτά σε άλλα κράτη-μέλη, όπως η Πολωνία, που δεν είναι τόσο πράσινη, που δεν έχει καθόλου τον ίδιο όγκο ανανεώσιμο όπως εμείς, τα ορυκτά καύσιμα που καταναλώνει παρόλα αυτά και που βλάπτουν το περιβάλλον αέριο φτάνει περίπου ε, στην περίπτωσή της κατά 66% από τη Ρωσία. Όμως έχει και δικά της ανθρακορυχία που βεβαίως δεν είναι καλά από την άποψη του διοξιδίου του άνθρακα αλλά ως προς την προμήθεια είναι ένα θετικό στοιχείο. Και άλλοι φίλοι όπως η Πολωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διαφορετικό βασικά αποθέματα σχιστολήθου Η Γαλλία αποφάσισε να μην αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Η Πολωνία ναι. Είναι κάτι που εξαρτάται από τους εμπορικές πατριώτες του καθενός, υποθέτω, αλλά η ερώτησή μου είναι αν σκεφτεί κανείς την ασφάλεια της παροχής, της προμήθειας. Πώς μπορεί να εξισορροπήσει τη μείωση των ε, εισαγωγών την ανάγκη της βιομηχανίας να έχει ανταγωνιστικές τιμές με την ανάγκη να επιτύχει κανείς τους στόχους που έχουμε θέσει για το κλίμα. Διότι σε κάποια κράτη-μέλη επιτυγχάνει κανείς τον ένα στόχο, αλλά φαίνεται να αντιφάσκει τελείως με τον άλλο. Είναι πολύ δύσκολη η εξισορρόπηση αυτών των τριών παραγόντων και στην Επιτροπή αυτή, στο Κοινοβούλιο, έχουμε περάσει την τελευταία πενταετία προσπαθώντα να δώσουμε έμφαση στην κλιματική διάσταση της ενέργειας, Σημαντικό, δεν το αρνούμε. Αλλά αν δούμε την ασφάλεια τη παροχή, προσκρούμε σε ε, προφανείς αντιφάσεις ε, ως προς τις ενεργειακές ανάγκες και τις ανάγκες του κόστους και το τι μπορούμε να κάνουμε πρόθεσμα Είπατε και προηγουμένως ότι οι ενενεώσιμες πηγές είναι πολύ σημαντικές στη χώρα μου με 33% όμως δεν μπορούμε να ε, ικανοποιήσουμε όλες τις ενεργειακές μας ανάγκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο συνάδελφος Νίκα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Pentru că cred că este cel puțin la fel de frumoasă ca și limba spaniolă. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα ρουμανικά είναι σχεδόν τόσο ωραία όσο τα ισπανικά, γι' αυτό και θα τα μιλήσω. Ε, κύριε Επίτροπε, έχετε ανάγκη από, ιταλική στήριξη, από ε, πολιτική στήριξη και θα την έχετε από πλευρά μα. Ε, δείξατε αποφασιστικότητα και ταχύτητα ε, στο να αντιμετωπίσετε τα διάφορα θέματα που σα έχουν ήδη τεθεί πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνήθως μάλλον, κατηγορείται για καθυστερήσεις ή για υπερβολική γραφειοκρατία. Ε, αυτό είναι το κλασικό επιχείρημα. Όμως ε, ε, εδώ ελπίζουμε να μας πείσετε για το αντίθετο. Και αυτό που πρέπει να πω είναι ότι εδώ χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα δράσης, πολύ συγκεκριμένο, και γι' αυτό ήθελα να μιλήσω για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ε, υπόθηκε και το γνωρίζουμε όλοι ότι ο μεγάλος όγκος της κατανάλωσης έχει να κάνει με την θέρμανση το χειμώνα και τον κλιματισμό το καλοκαίρι στην Ευρώπη. Όμως η έγκριση της οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα είναι επίγουσα. Εάν το 30% των ε, λογαριασμών ε, της ενέργειας ήταν φθηνότερο από το 30% που καταναλώνουμε, ξέρουμε τι αντικτύπωση θα υπήρχε για τους πολίτες μας. Δεν ε, θα ήταν πολύ καλό να μπορούμε όντως να ελέγξουμε έτσι την κατανάλωση. Αλλά εάν η παραγωγή χάλιβα λόγω χάρη μπορούσε να παραμένει στην Ευρώπη διότι δεν θα κατανάλωνε πολύ ενέργεια. Δεν θα ήταν και αυτό πολύ ευχάριστο. Η ενέργεια λοιπόν πρέπει να παράγεται με τρόπο ανταγωνιστικό αλλά προς με σεβασμό προς, όλες τις, προς όλους τους περιβαλλοντικούς και οικολογικούς μας κανόνες. Πέραν αυτού, είναι σαφές ότι χρειάζονται επενδύσει για την έρευνα. Ε, αναφέρατε δύο πτυχές που τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Πρώτα απ' όλα η αυτοκινητοβιομηχανία. τα ε, αυτοκίνητα δεν είναι πλέον τόσο δημοφιλή στην Ευρώπη. Διότι τα ηλεκτρικά οχήματα εννοώ είναι, δεν είναι τόσο δημοφιλή ακόμα στην Ευρώπη διότι δεν υπάρχει σύστημα αναφοδιασμού. Δεν ξέρει κανεί πού να κάνει τη φόρτιση. Ε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να επιληθεί. Ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε λοιπόν εδώ να είναι καθοριστικό ή για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε δύο πτυχέ. Κατά πρώτον, η τιμή πώληση τη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από, και, από ηλιακέ και ολικέ πηγέ δεν νομίζω ότι είναι όρθη. Πολλέ φορέ είναι, είναι πολύ ψηλή η τιμή αυτή τη ενέργεια. Αυτό ίσω δεν έπρεπε να είναι έτσι. Και αν με την έρευνα πετυχαίναμε να περιορίσουμε αυτές τις τιμές, να τις ελέγξουμε, θα ήταν πολύ ωραίο. Αλλά η τιμές ε, της ενέργειας που προκύπτουν από αυτές τις πηγές είναι πολύ υπερτιμημένες. Πολύ περισσότερο και από τα ορυκτά καύσιμα. Εάν δείξετε ότι είστε ταχύς όμως στις αποφάσεις σας, θα έχετε όλη την απαραίτητη πολιτική στήριξη και για θέματα που δεν αναφέρθηκαν ενδεχομένω. Αν και ε, σχολιάσετε πολλέ από τι δικέ μα ανησυχίε. Ευχαριστούμε εκ μέρου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριο Αλέκοφ. I speak my uh, Θα μιλήσω και εγώ τα βουλγαρικά, τη μητρική μου γλώσσα. Γεια σας. Να χαιρετήσουμε τον ε, προσκεκλημένο μας, τον κύριο Επίτροπο. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας. Και να επανέλθω στα όσα αναφέρετε. Μου έκανε Μα έκανε εντύπωση η αντίδραση του κυρίου Πούτιν. Ε, ήταν έκπληξη η αντίδραση τη Ρωσία για του συναδέλφου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για του βουλγάρους ε, συναδέλφου. Μα εξέπληξε το γεγονό ότι η Ρωσία σκοπεύει να σταματήσει τα σχέδιά τη για τον νότιο αγωγό. Σήμερα ακούσαμε ότι δεν είναι αξιόπιστος τέλο η Ρωσία για την προμήθεια ενέργειας στην Ευρώπη. Θα ήθελα να αναφέρω ότι σας ευχαριστώ για το θέμα που αναφέρατε σχετικά με την σταθερότητα την ενεργειακή στην Ευρώπη. Και εδώ λοιπόν έρχεται το ερώτημά μου. Ποια είναι η ευρωπαϊκή μας στρατηγική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντισταθμίσουμε την έλλειψη και την ανάγκη ενέργειας ως απόρρια του τερματισμού του έργου αυτού. Ποια είναι η θέση μας σε ό,τι αφορά τον νότιο αγωγό, ποιες είναι οι εναλλακτικέ λύσεις για την συνέχιση ενδεχομένως κάποιων τμήματων του έργου αυτού. Γιατί σήμερα έγιναν δηλώσεις από τον συνάδελφό σας κύριο Σεύκοβιτς ότι προτίθεται ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποια συνέχιση. Ε, υπάρχει κίνδυνος μονομερός να αποφασίσει ο κύριος Πούτιν σε ό,τι αφορά τον αγωγό που περνάει από την Τουρκία και από τη Βουλγαρία που είναι το δεύτερο πιο νότιο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και μπορείτε να υπολογίσετε στην υποστήριξή μας ότι αφορά θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Ευχαριστώ ο συνάδελφος Βιντάλλα. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμε κύριε Καρίες Κανιέτε. Την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Γιούγκερ παρουσίασε το επενδυτικό του σχέδιο που υποτίθεται ότι θα εξυπηρετήσει την ευρωπαϊκή οικονομία διότι θα διεγείρει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Σίγουρα λείπουν επενδύσεις από την Ευρώπη γιατί υπάρχουν πολλές αγκυλώσεις και οι ανταγωνιστές μας απ' την άλλη δεν έχουν καμία αγκύλωση αλλά άρα πολύ δυναμισμό. Και αναφέρομαι ε, και στους παραδοσιακούς ανταγωνιστές μας και στις αναδυόμενες οικονομίες. Και γι' αυτό πολλοί επίτροποι θέλουν ε, το σχέδιο επενδύσεων του Προέδρου Γιούνκερ να το τραβήξουν προς το δικό τους χαρτοφυλάκιο. Θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε ένα μέρος των 300 δις που υπάρχει ελπίδα να κινητοποιηθούν για να έχουμε μια πιο ανταγωνιστική ενέργεια. Είναι πολύ γνωστό ότι όταν μειώνεται το τιμολόγιο της ενέργειας βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας και δημιουργούνται περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Με δεδομένη την οικονομική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η Ευρώπη, η προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι ε, ε, η ενέργεια να είναι εφικτή να είναι προσβάσιμη για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες. Και ένας τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι να ε, ε, υλοποιήσουμε μια πραγματική εσωτερική ενιαία αγορά ενέργειας και ο στόχος αυτός χρειάζεται συνένεση. Πολλά έχουν γίνει σε αυτό το πεδίο, το αναγνωρίζω. Ωστόσο τα κενά είναι επίσης πολλά και μεγάλα. Το πιο πασιφανές παράδειγμα, οι ενεργειακές νησίδες. Δεν μπορούμε να μιλούμε για ενιαία αγορά ενέργειας όταν σε κράτη ε, ε, υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν είναι διασυνδεδεμένα με τις υπόλοιπες, π.χ. η Βυρική Χερσόνησος, οι χώρες της Βαλτικής. Σας ερωτώ λοιπόν, έχετε μελετήσει προς τα πού θα κατευθύνετε τις επενδύσεις, θα χρηματοδοτήσετε σχέδια διασύνδεσης μεταξύ των χωρών μελών. Άλλο μεγάλο μέλημα της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής είναι η βελτίωση του οικονομικού κλίματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οποίες είναι και το 99% του επιχειρηματικού ιστού στην Ευρώπη, του εργοδοτικού ιστού στην Ευρώπη. Σε αυτές οφείλουμε τα δύο τρίτα των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να σας φαίνεται ε, περίεργο κύριε Επίτροπε, αλλά επιτρέψτε μου να αναφερθώ στις μικρομισές επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας. Είναι δύσκολο να τις εμπλέξουμε. Το δέχομαι, αλλά δεν είναι ανέφικτο. Κοιτάξτε, οι μεγάλοι εργολάβοι, οι μεγάλοι ανάδοχοι αν θέλετε, πρέπει να αναλάβουν και τις μεγάλες ευθύνες, γιατί παίρνουν και τα πιο μεγάλα συμβόλαια. Μπορεί κανείς να κάνει λόγο για τεράστιες υποδομές και καλώς. Ας μιλήσουμε όμως ότι σε όλους τους οικονομικούς κλάδους υπάρχει κάποιο αφεντικό. Και όχι μόνο κάποιο αφεντικό, υπάρχει κάποιος καθοδηγητής, αλλά υπάρχει και κάποιο μοντέλο, υπάρχει και κάποιο πρότυπο. Ε, όλα για να γίνει κάποιος μεγάλος έχει ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μοντέλο, έχει ένα συγκεκριμένο πρότυπο, έχει κάνει καινοτομίε, έχει επινοήσει πράγματα και όλα αυτά υπάρχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ξέρετε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις κάνουν outsourcing, εξωτερικεύουν, αναθέτουν σε εξωτερικούς συμβούλους και πρέπει ε, να το γνωρίζουμε και εμείς αυτό, να πιάνουμε, να συλλαμβάνουμε το πνεύμα των καιρών και θα πρέπει να αναγνωρίζουμε την διαφάνεια, την εντιμότητα αλλά και την διαδρομή, τα προηγούμενα όλων αυτών των αναδόχων, τα καλά και τα κακά. Κλείνω λέγοντας ότι αναφερθήκατε στο στόχο ε, σταθεροποίησης της προμήθευσης σε ενέργεια ε, με δεδομένο ότι έχει εγκαταλειφθεί η ιδέα του South Stream. Θα ήθελα να γνωρίζω το εξής. Και ξέρω ότι δεν το είπατε για να σημάνετε το ο καμπανάκι του συναγερμού, αλλά αφού θέλετε να μας καθησυχάσετε, ίσως θα πρέπει εμείς να ανησυχήσουμε λίγο και γι' αυτό θέτω το εξής ερώτημα. Ποιες νομίζετε ότι θα είναι οι συνέπειες της απόφασης που έλαβαν οι ρωσικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Γιαβόρα από τους Πρασίνους. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε και να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Κύριε Επίτροπε, αναφέρετε ότι έγινε ένα περιστατικό στην μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ουκρανία, στην Νότιο Αυχαζία. Θα, μπορούτε να, θα μπορούσατε να μας δώσετε πληροφορίες στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Ήτρε, κάποιες πληροφορίες πέρα από τις πληροφορίες που δίνουν τα μέσα ενημέρωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιπρόσθετες πληροφορίες για ενδεχόμενη ρήπανση ή οποιοδήποτε τέτοιο πυρηνικό περιστατικό στο εργοστάσιο αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε και τώρα εξ ονόματος ε, της ΓΚΟΕ, η κυρία Λόμπες Πριμέγιο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε, θα ήθελα να αδράξω αυτή την ευκαιρία, αυτό το διάλογο, για να σχολιάσω το πρόβλημα των βιομηχανιών υψηλής εντάσεως ενέργειας, όπως είναι ο κλάδος της μεταλλουργίας. Την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια σχολιάζαμε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χαλιβουργία στο Τέρμι, στην Ιταλία. Και δυστυχώς αυτή τη εβδομάδα αναγκαστήκαμε να μάθουμε την ε, δραματική η κατάσταση της επιχείρησης Αλκόα, της ισπανικής επιχείρησης, ε, που μια επιχείρηση που είναι στη δική μου και στη δική σας χώρα και από αυτήν εξαρτώνται Τοντάδε άμεσε θέσεις απασχόληση και χιλιάδε έμεσε θέσει απασχόληση σε μια ζώνη πάρα πολύ προβληματική από πλευρά οικονομική όπω είναι η περιοχή τη Αστούρια. Η μετεγκατάσταση τη Ευρωπαϊκή ε- Βιομηχανία σε άλλε χώρε αποτελεί μεγάλη απώλεια για την απασχόληση και τον ευρωπαϊκό βιομηχανικό ε, ιστό. Είναι μια απώλεια που επηρεάζει τη ε, δουλειά αυτή τη επιτροπή, διότι η βιομηχανία που χάνουμε είναι η πιο αποτελεσματική από πλευρά εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και από άλλων ρήπων. Στηρίζουμε λοιπόν μια φιλόδοξη στρατηγική ε, περιβαλλοντική αποδοτικότητα και θα πρέπει αυτή να συμβαδίζει με συμπληρωματική στρατηγική έτσι ώστε να έχουμε οικολογικά πρότυπα ίδια για τι εισαγωγέ που κάνουμε. Και όχι μόνο αυτά, η ενεργειακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση απελευθέρωσε ένα κλάδο, τον ηλεκτρικό κλάδο, το κλάδο τη ηλεκτρική ενέργεια, ο οποίο εκφύσεως ήταν ένα κλάδο με ολιγοπόλια ιδιωτικά. Γνωρίζετε πολύ καλά την κατάσταση στην Ισπανία. Ήσασταν συνένοχος της κυβέρνησης ε, όταν έκανε αυτή την ανεπαρκή ε, κανονιστική ρύθμιση, όταν νομοθετούσε ε, με ανεπαρκή, ανεπαρκή τρόπο. Έχει συγκεντρωθεί σε πολύ λίγους φορείς εκμετάλλευσης όλη αυτή η δυνατότητα, όλη αυτή η εξουσία και αυτό πλήττει τους πολίτες και την παραγωγική οικονομία. Και αυτό σπρώχνει την Αλκόα και την Τίσεν να κλείσουν. Δεν υπάρχουν τιμολόγια βιομηχανικά, δεν υπάρχει σύστημα ρύθμισης των ολιγοπολίων στοιχείων δεν, δεν θέλουμε να φτηνίνει η ενέργεια γιατί θα έχουμε προσφύγει σε επικίνδυνες τεχνολογίες όπως είναι η πυριανική ενέργεια ή η υδροροκμάτωση. Θέλουμε η υδροροκματεωση θελουμε η ενεργεια να ξαναπεράσει στον έλεγχο του δημοσίου, να προσαρμόσουμε το σύστημα των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στις ανάγκες ενός διαφοροποιημένου παραγωγικού μοντέλου το οποίο δεν θα παρετείται από τη βιομηχανική του βάση. Και γι' αυτό δεν μας ταιριάζει η ενεργειακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντί να δρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ανακτήσει τον έλεγχο ενός στρατηγικού επιχειρηματικού κλάδου παρουσιάζει ένα πρόγραμμα μεγάλων υποδομών και ε, ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Υπήρου και έτσι η ηλεκτρική αγορά θα συγκεντρωθεί ακόμα περισσότερο στα χέρια ολίγων και έτσι η Ευρώπη θα είναι συνένοχο στην απώλεια χιλιάδων θέσεων απασχόλησης ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Ταμπουράνο, εξ ΕΕ. Ε, γεια σας, Επίτροπε Κανιέτε. Ε, σας ευχαριστούμε και για την εισηγησή σας, αλλά ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία που μου φαίνονται πιο ενδιαφέροντα. Ε, το σύστημα ανταλλαγής εκπομπών αερίων, δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οικολογικά σήματα και γενικότερα τα, η ετικετοθεσία, η επίθεση ετικετών. πρέπει η επισήμανση μάλλον. Για το ETS πρώτα απ' όλα λοιπόν, το σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων οριών του θερμοκηπίου. Είδαμε ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση διότι δεν λειτουργεί. Έχει γίνει ένα μέσο κερδοσκοπίας για το διεθνές εμπόριο και καθόλου δεν λειτουργήσε όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Στον ε, ΠΟΕ άλλωστε έχουν καταφέρει αυτοί που ε, ενδιαφέρονται να το χειριστούν το σύστημα αυτό να το μετατοπίσουν εκεί που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να είναι αποτελεσματικό το ETS. Είναι ίσως ε, περίεργο ένα μέλος της Επιτροπής αυτής που έχει οικολογικές ανησυχίες να ζητά την κατάργηση του συστήματος ETS και καλύτερα να υπήρχε ένας φόρος για τον άνθρακα όπου να υπολογίζεται το περιεχόμενο η περιεκτικότητα σε διοξίδιο του άνθρακα ανάλογα με τα προϊόντα που καταναλώνονται. Προϊόντα όμως που έχουν παραχθεί. Δεν είναι μέτρο προστατευτισμού, απλώς θα έπρεπε να ε, επιτρέψει στην ε, διεθνή αγορά μάλλον να επιτρέψει αυτό το μέτρο στην ευρωπαϊκή αγορά να ανταγωνιστεί με ίσους όρους στη διεθνή αγορά και όχι ξένα προϊόντα να φτάνουν στην επικράτειά μας ε, με αθέμητο ανταγωνισμό και πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Θα συνεργαστώ με περίπου ε, ε, με μια ομάδα Ιταλών ερευνητών που θα προτείνει αυτή την πρωτοβουλία για τον συγκεκριμένο φόρο. Σας ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε. Μετά τις παρεμβάσεις των ε, συντονιστών μας, να ζητήσω από τον Επίτροπο να απαντήσει. Mm. Ευχαριστώ πολύ. Μου τέθηκε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα η κατάσταση των διαφόρων χωρών μελών είναι πολύ διαφορετική από πλευράς επάρκειας στην προμήθευση ε, ενέργειας. Άλλα κράτη είναι εξαιρετικά εξαρτώμενα, σε άλλα κράτη έχει μεγάλο βάρος ε, όλος ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, άλλα εξαρτώνται πολύ περισσότερο από τρίτες χώρες. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς λοιπόν για να εγγυηθούμε ότι τα κράτη-μέλη θα είναι πιο ανταγωνιστικά. Πιστεύω ότι το πρώτο που πρέπει και μπορούμε να κάνουμε είναι να ε, φροντίσουμε για όλες τις απαραίτητες διασυνδέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσουμε όλα αυτά τα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και συμφέροντος, να εγγυηθούμε ότι θα έχουμε μια ενιαία, μοναδική, πραγματική, εσωτερική ενέργεια, όπου θα κυκλοφορεί και το φυσικό αέριο και τα νεώσιμες πηγές, ε, το πετρέλαιο, όλες οι πηγές ενέργειας θα κυκλοφορούν απρόσκοπτα. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να καταπολεμήσουμε τα μονοπόλια στην προμήθευση και πρέπει καταπολεμήσουμε και την εξάρτησή μας από έναν και μοναδικό προμηθευτή. Το είδαμε και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Τι πρόβλημα δημιουργείται όταν κλείνει η στρόφιγγα για το φυσικό αέριο σε μια χώρα. Μπορεί να... Ε, να ε, καταπνιγεί η οικονομία της χώρας αυτής και να καταδικαστούν οι κάτοικοι σε μια ε, ζωή η οποία θα είναι κόλαση. Γι' αυτό θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε λοιπόν τους προμηθευτές μας. Χρειαζόμαστε ε, ε, δίκτυο υγροποιημένου φυσικού αερίου το οποίο να μας επιτρέπει να έχουμε εναλλακτικέ. Έχουμε εξαρτηθεί πάρα πολύ από το φυσικό αέριο ε, ρωσικής προέλευσης. Πρέπει να εξαρτηθούμε περισσότερο αν θέλετε από το φυσικό αέριο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και πρέπει να έχουμε μια πραγματική ολοκληρωμένη ενιαία ενεργειακή αγορά και για να το καταφέρουμε αυτό πρέπει να δουλέψουμε πρώτον στις υποδομές, δεύτερον στον τομέα των network codes για να είναι διαλειτουργικά τα δίκτυα. Πρέπει να δουλέψουμε στο επίπεδο της περιφερειακής συνεργασίας, η οποία έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Αλλά δεν αρκεί να λειτουργεί καλά μόνο η περιφερειακή συνεργασία σε δύο-τρία σημεία της κεντρικής Ευρώπης π.χ. ή στις χώρες της Βαλτικής. Πρέπει να είναι πραγματικά όλη η ευρωπαϊκή αγορά ενία και πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι διαδικασίες για, τη, ε, για τον καθορισμό των τιμών να είναι πολύ πιο διαφανείς. Κατανοώ ε, την παρέμβαση της εκπροσώπου ε, της πολιτικής ομάδας της, αριστερά, της αριστεράς. Δεν είναι το πρόβλημα το μονοπόλιο της ΧΕΨΗ εταιρεία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μια αγορά όπου να ανταγωνίζονται η μία την άλλη ε, ε αυτές οι εταιρείε. Και γι' αυτό πρέπει να φτιάξουμε μια... Ε, ενιαία αγορά όπου οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και έτσι θα ωφεληθεί ο καταναλωτής. Και αν υπάρχει μονοπόλιο, λιγοπόλιο σε μια χώρα, 7 εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλη χώρα, σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε μια ενιαία περιοχή, έναν ενιαίο χώρο, απτό χώρο, φυσικό χώρο όπου όλες οι εταιρείες θα είναι ανταγωνιστικές, τότε θα έχουμε αποτέλεσμα για το καταναλωτή και θα υπάρχει επάρκεια στην προμήθευση. Είναι φιλόδοξο το σχέδιό μας, έχουμε προχωρήσει πολύ και πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν καταρτήσουμε τα συστήματα διακυβέρνησης θα πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε αυτά να είναι ευέλικτα, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική κατάσταση του εκάστοτε κράτους μέλους. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να έχουν όλα τους ίδιους ταυτόσιμους στόχους πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που έχουν να αναπτύξουν τη χή υψή μορφή ενέργειας. Χαίρομαι και ε, ευχαριστώ τον εκπρόσωπο των ε, σοσιαλιστών για την πολιτική στήριξη που μου προσέφερε, την οποία και θα χρειαστώ για τη δουλειά που καλούμε να κάνω σε αυτό το πεδίο. Λέω ότι συμφωνώ μαζί σας, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πολύ προσεκτική και να είναι επιμελής στα καθήκοντά της. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στις 30 μέρες που είμαι επίτροπες, ε, επί 30 μέρες που είμαι επίτροπος, όλη η Επιτροπή εργάζεται με εντατικού ρυθμούς. Έχουμε παρουσιάσει το σχέδιο Juncker, έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα εργασιών, δουλεύουμε πάνω στην ημερήσια διάταξη με πολύ μεγάλη ταχύτητα, δηλαδή η μηχανή δουλεύει στο φουλ γιατί επήγει το ζήτημα, επήγουν όλα τα ζητήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Μίλησε λοιπόν για την ενεργειακή επάρκεια και για τη δυνατότητα αναθεώρησης της σχετικής οδηγίας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η οδηγία είναι καλή και καλώς υπάρχει. Ενδεχομένως δεν την έχουμε εφαρμόσει επαρκώς. Όταν έχουμε περιπτώσεις μη ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο ή μερικής ενσωμάτωσης των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και αναφέρομαι εδώ σε 13 ή 14 κρατημέλη όταν βλέπουμε 20 ε, πιλωτικά σχέδια και 20 ε, χώρες μέλη είναι σε πιλωτικό στάδιο ακόμα ε, όλο αυτό σημαίνει ότι δεν την έχουμε υλοποιήσει 100% για να αναθεωρήσουμε μια οδηγία πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζεται όταν έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωσή της 100% ας εφαρμοστεί πρώτα να δούμε πώς εφαρμόζεται και να αναθεωρούμε μετά εάν θεωρείτε ότι κάποια πτυχή της οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα ε, είναι λυπές, κάποια, είναι ε, λυπής κάποια πτυχή, να μου το διαβιβάσετε. Τα μηνύματα που λαμβάνω εγώ είναι ότι είναι καλή η οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα, ότι έχει γίνει πολλή δουλειά και ότι εάν εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Στον κύριο Μπάρεγκοφ στρέφομαι τώρα για να πω το εξής. Μιλήσατε για το... για το τι θα κάνουμε ε, μετά τις ε, ε, τελευταίες αποφάσεις των ρωσικών αρχών και του Προέδρου Πούτιν, ο οποίος αποφάσισε την ακύρωση του έργου για το South Stream. Η Επιτροπή λοιπόν επαναλαμβάνει ότι καταγράφει την λήψη αυτή, ε, της, αυτής της μονομερούς απόφασης και ότι θα αξιολογήσει την κατάσταση. Η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν θεωρούσε ότι ο South Stream δεν είναι ένα έργο το οποίο θα αυξήσει την ασφάλεια της ε, ε, προμήθευσης της ενέργειας στην Ευρώπη. Το μόνο που θα έκανε ήταν να δώσει μια εναλλακτική δίωδο, έναν εναλλακτικό αγωγό μέσω του οποίου θα έρχεται η ενέργεια στην Ευρώπη. Αλλά δεν βοηθάει στο να μην έχουμε ένα μόνο προμηθευτή και στο να διαφοροποιήσουμε τις πηγές μας προμήθευσης. Επομένως, η κατασκευή, η λειτουργία του South Stream πρέπει να συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο, με ε, τους κοινοτικούς κανόνες για τις ε, δημόσιες αγορές, για τους δια, διαγωνισμούς, ε, για την πρόσβαση στο διαγωνισμό, για τη συμμετοχή, για τον τρόπο με τον οποίο θα κατασκευαστεί και το καθεξής. Ε, τι συμβαίνει. Ε, αυτό το οποίο υπόθηκε είναι ότι με τις υφιστάμενες συνθήκες σταματάει το έργο. Εάν οι ρωσικές αρχές δεχθούν το κοινοτικό δίκαιο και την εφαρμογή του σε αυτή την περίπτωση, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συνεχίσουμε ε, με το South Stream. Όμως όλα αυτά συζητούνται ε, το τρίτο πακέτο ενέργειας στο πλαίσιο του ΠΟΕ αυτή τη στιγμή. Ε, αν δεν υλοποιηθεί ο South Stream, πώς θα έχουμε σίγουρη προμήθεια σε ενέργειες, σε πηγές ενέργειας ε, στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να επιτεχύνει τις εργασίες της έτσι ώστε αυτές οι περιφέρειες να συνδεθούν όσο δυνατόν νωρίτερα και γρηγορότερα με την υπόλοιπη Ευρώπη από πλευράς δικτύων ενέργειας. Έχουμε τον αγωγό που θα συνδέσει Βουλγαρία-Ρουμανία, αυτό που θα συνδέσει Βουλγαρία-Ελλάδα ή τον κεντρικό διάδρομο που περνάει από τη Ρουμανία και ούτε καθεξής. Πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια, πρέπει να υλοποιήσουμε αυτά τα έργα το συντομότερο δυνατόν για να εγγυηθούμε τον εφοδιασμό αυτών των περιοχών. Θα υπάρξει συνάντηση με τους Αμερικανούς συναδέλφους στο πλαίσιο της μόνιμης συνεργασίας που έχουμε για ενεργειακά ζητήματα θα ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε για να στηρίξουμε όλα αυτά τα έργα κοινωνικού, κοινοτικού με ενδιαφέροντος. Μιλήσατε επίσης για τις ενεργειακές νησίδες και εμείς θα παρουσιάσουμε ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εφαρμόζει τη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Να έχουμε 10% διασύνδεση το 2020 και 15% διασύνδεση το 2030. Στη συνέχεια όμως αναφερθήκατε ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο πόσο θα πρέπει να τις στηρίξουμε και θέσατε και σχετικό ερώτημα κατά πόσο μπορούμε να πάρουμε κάποια κονδύλια από το σχέδιο Juncker για να το αφιερώσουμε σε ε, υποδομές για τις διασυνδέσεις. Και λέγοντας ότι πράγματι, διαβάζοντας το σχέδιο Juncker, βλέπουμε ότι προτεραιότητα θα έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι επενδύσεις σε υποδομές διασύνδεσης και ενεργειακή αποδοτικότητα. Το πεδίο της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι πολύ σημαντικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Γρήγορα δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης σε αυτό το τομέα. Τα έργα υποδομής για να οριμάσουν χρειάζονται δύο ή τέσσερα χρόνια ή και πέντε, γιατί πρέπει κανείς να έχει περιβαλλοντικές άδειες, διοικητικές άδειες, ε, πρέπει να γίνουν πολλά και διάφορα. Η ενεργειακή αποδοτικότητα όμως, δηλαδή το να δουλέψει κανείς πάνω σε κτίρια, δημόσια ή ιδιωτικά, είναι κάτι που μπορεί να κάνει αμέσως. Επομένως, εάν αρχίσει να εφαρμόζεται με το ε, σχέδιο Juncker αριθμός φιλόδοξων προγραμμάτων ε, πάνω στο πεδίο και στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας θα έχουμε άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης και έτσι θα κινητοποιηθούν και κεφάλαια και θα υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό βάση ε, του σχεδίου Juncker 75 δις θα διοχετευτούν προς αυτή την κατεύθυνση από τα 315 επομένω ε, σε 75 δις διοχετεύονται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λαμβάνουμε υπόψη τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, την ενεργειακή αποδοτικότητα. Είναι αλήθεια ότι η μικρομεσαία επιχειρήση δεν θα μπορέσει να συμβάλλει π.χ. στις μεγάλες υποθαλάσσιες διασυνδέσεις, κάτι το οποίο, ε, ε, για το οποίο είναι πιο κατάλληλες οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Μπορούν όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμβάλλουν, να δουλέψουν π.χ. στα συστήματα θέρμασης, ψήξης σπιτιών με μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα σε τέτοιου είδους μικρής κλίμακας έργα ε, σε τέτοιου είδους έργα μικρής κλίμακας στο δημόσιο ή το ιδιωτικό τομέα. Ε, βάσει των στοιχείων που έχουμε αυτή τη στιγμή από την Ευρατόμ, έχουμε ένα, πρόβλημα στο μετασχηματιστή, στην τρίτη μονάδα ε, πυρηνικού αντιδραστήρα στην Ουκρανία. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις. Ε, επισκευάζεται η βλάβη αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία και θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία το σύστημα στις 7 Δεκεμβρίου. Δεν έχουν καταγραφεί μη φυσιολογικά επίπεδα ραδιενέργειας στην ε, EURDEP που είναι η αρμόδια υπηρεσία που παρακολουθεί όλα όλα αυτά και ούτε υπάρχει ε, πρόβλημα με το σύστημα EQRE e, όπου σημαίνεται το καμπανάκι του συναγερμού για θέματα πυρηνικής ενέργειας. Όλες μας οι επαφές, οι επίσημες επαφές μας λένε λοιπόν ότι ε, όλα είναι στα φυσιολογικά επίπεδα, η βλάβη επισκευάζεται, δεν έχει περαιτέρω επιπτώσεις. Το συμβάν ε, καταχωρίζεται ε, στη ζώνη μηδέν της κλίμακας επικινδυνότητας και ε, γρήγορα θα υπάρξει σχετική έκθεση η οποία θα επιβεβαιώσει ε, αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό είναι το μέγεθος, το βεληνικές αν θέλετε, του συμβάντος ε, του προβλήματος ηλεκτρικής βλάβης στον συγκεκριμένο αντιδραστήρα στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα, άλλος ε, συνάδελφός σας αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό και στην αγορά. και μίλησε για τις βιομηχανίες υψηλής εντάσεως ενέργειας. Η συνάδελφός σας λοιπόν μοιράστηκε μαζί μας ε, τις ανησυχίες της ε, με τις οποίες συμφωνούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Βράχει πρόθεσμα. Λαμβάνουμε υπόψη μας τέτοιου είδους βιομηχανίες κατά την κατανομή το, στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, ρήπων, σε κάθε περίπτωση η πολιτική μας έχει ως στόχο να φτηνίνει το τιμολόγιο ενέργειας και αν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης τότε μειώνεται ο λογαριασμός για τη βιομηχανία και για τους πολίτες. Όσο περισσότερη διαφοροποίηση έχουμε τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να μειώσουμε το κόστος και τόσο πιο ανταγωνιστικοί θα γίνουμε. Επομένως, ό,τι κάνουμε έχει να κάνει με την αναζήτηση ενός πιο αηφόρου συστήματος με πιο φτηνή ενέργεια και αυτό επιτυχάνεται με την πραγματικά ενιαία αγορά ενέργειας. Αν ενισχύσουμε την αγοραστική δύναμη και αυτό μελετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν εκπληρωθούν ορισμένες ε, κανονιστικές διατάξεις εφαρμοστούν, δουλεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση συγκεκριμένες παραδοχές. Αν μπορούν κάποιε εταιρείε να ενωθούν για να ενισχύσουν την αγοραστική τους δύναμη, ε, έτσι θα υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες ε, στους διαγωνισμούς και στην ανάληψη των έργων. Ε, ασκήθηκε επίσης κριτική στο σύστημα εμπορίας ρήπων. Ε, όταν εξετάσαμε όλες αυτές τις ε, επιλογές για το πώς θα πετύχουμε τους στόχους έτσι ώστε η οικονομία μας να εξαρτάται όλο και λιγότερο από το ανάνθρακα, τέθηκε αυτό το πρόβλημα του carbon tax, αυτού του φόρου. Έχει πάρα πολλά ελαττώματα αυτό το σύστημα, σας το εξήγησα στην ακρόαση. Θέλουμε το σύστημα εμπορίας ρήπων να βελτιωθεί, να γίνουν τροποποιήσεις οι οποίες γίνονται σιγά σιγά, να λειτουργήσει και τελικά να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα μας επιτρέψει να απομακρυνθούμε από μια οικονομία που θα βασίζεται ε, στον άνθρακα, αλλά θα έχουμε σωστή κατανομή του ε, συνεπαγόμενου βάρους σε όλους τους φορείς. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος για τον επόμενο γύρο ερωτήσεων και πατρίσεων. Ο συνάδελφος Πέτερλε, λοιπόν. σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Επιτροπή Καλνιέτε, που βρίσκεστε μαζί σα σήμερα. Κύριε Πέντερλε, να σα πω ότι από πλευρά τη ομάδα μα μα ανησυχούν οι φήμε για τη λίστα του Juncker, ε, η λίστα μεταρρύθμιση, όπω αναφέρεται στου κόλπου τη Επιτροπή ενδεχομένω του Γιούγκερ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πακέτο για τη διαχείριση τη ποιότητα του αέρα της ατμόσφαιρας. Υπάρχουν κάποιες φήμες που λένε ότι θα καταργηθεί την επόμενη εβδομάδα. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε τις εργασίες αυτές στο Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το MCP, επί του οποίου εργαζόμαστε στην παρούσα φάση. Είμαι εισηγητής από την Επιτροπή Ήτρα για το θέμα αυτό. Θα ήθελα το συντομότερο δυνατόν να γνωρίζω αν θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και το τι συμβαίνει γενικότερα. Είναι πολύ σημαντική η εργασία μας, ξέρετε, και για το περιβάλλον και για την υγεία. Επίσης, πέρα από τους στόχους για το 2030, ε, αναρωτιέμαι θα υπάρξουν νομοθετικές προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου για να εφαρμοστούν σιγά σιγά οι στόχοι που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που έχουν επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα ζητήματα αυτά και στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Μπρέμπτ. Bremt. Ναι, Φανμπρέμπτ διορθώνει. Να σας ρωτήσω, κύριε Επίτροπε, το εξής. Συγκεκριμένες ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Καταρχάς, αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας το γεγονός ότι του χρόνου θα κάνετε μελέτη αντικτύπου α, για το μη ETS. Έχω κάποιες ανησυχίες. Έχει ξεκινήσει η Σύνοδο στη Λίμα, προετοιμαζόμαστε για το Παρίσι και εδώ στο Κοινοβούλιο λέμε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέτουμε το καλό παράδειγμα, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος, γιατί αυτό θα μας καταστήσει πιο δυνατούς εταίρους στις διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά και τις άλλες περιφέρειες και περιοχές του κόσμου. Είναι λοιπόν θεωρώ πολύ σημαντικό να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για το ETS και για τομεί που δεν εντάσσονται στο ETS, στο σύστημα εμπορία ρήπων, όπω οι μεταφορέ. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει αυτό και να μην απαντήσουμε υπερβολικά πολύ χρόνο σε μελέτε αντικτύπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το αποφασίσει αυτό. Δεύτερη ερώτηση και πάλι για το κλίμα. Σε ό,τι αφορά τη Λίμα και το Παρίσι, αλλά καταρχάς σε ό,τι αφορά τη Λίμα. Δεν έχουν ανταποκριθεί όλα τα κράτη-μέλη έως σήμερα σε ό,τι αφορά τη διάθεση πόρων για το κλίμα και για το περιβάλλον, όπως η Αυστρία, όπως το Βέλγιο. Αυτό πραγματικά είναι ντροπή και μας ε, αποδυναμώνει ως εταίρους στη διαπραγματεύσεις. Ρωτώ λοιπόν, Επίτροπε, τι θα κάνετε για τις χώρες εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά το Ταμείο για το κλίμα. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα το πράξουν αυτό χώρες όπως η Αυστρία αλλά και το Βέλγιο, το συντομότερο δυνατόν μάλιστα. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Φαμπρέμπτ. Κύριε Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για την εισήγησή σας, Επιτροπέ. Μετάβαση για την απαλλαγή της εξάρτησης από τον άνθρακα στην οικονομία μας. Πολύ μεγάλης σημασίας Πρέπει να δούμε πώς σκοπεύει αυτή τη μετάβαση να την υλοποιήσει η Επιτροπή. Το λέμε ήδη από τη Σύνοδο του Κανκούν και για την ώρα δεν έχουμε δει να κάνει τίποτα σχετικά η Επιτροπή. Όλα τα μέτρα για την περιορισμό του κόστους, όπως την ε, κράτηση και την αποθήκευση άνθρακα. Αυτά χρειάζονται κέρυε τεχνολογικέ κινήσει και μένουμε πίσω παρόλα αυτά. Μένω σε μια περιοχή όπου δεκάδες χιλιάδες ε, θέσεις εργασίας εξαρτώνται από ε, την ε, ενέργεια ενέργειες που χρειάζονται, βιομηχανία που χρειάζεται μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Οπότε μας απασχολεί ιδιαίτερως η αποθήκευση και κράτηση άνθρακα. Εδώ στη Βόρεια Θάλασσα πρέπει να σκεφτούμε τον ιδιαίτερο ρόλο που υπάρχει και τις δυνατότητες μεταφοράς αποθηκευμένου άνθρακα, αλλά και τη δυνατότητα χάραξης νέων προγραμμάτων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Τούρμας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε για την ευρία επισκόπηση. Ήθελα να πω το εξή. Η συζήτηση για την ενεργειακή επάρκεια, την ενεργειακή ασφάλεια. Δεν συμφωνώ με την ε, ανάλυση του κυρίου Καρίνς. Δεν είναι πρόβλημα του τομέα της ενέργειας. Είναι πρόβλημα του τομέα της θέρμανσης. Δεν είναι τα εργοστάσια υπεύθυνα. Ε, έχουμε λιγότερο αέριο για τα εργοστάσια όσο ποτέ τα τελευταία δέκα χρόνια. Γιατί, γιατί με το ETS δόθηκε έμφαση στο αέριο. Το πρόβλημα της Ανατολικής Ευρώπης λοιπόν με τον κύριο Πούτιν είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να παγώσουν στα σπίτια τους μέσα. Γιατί τα κεντρικά συστήματα θέρμανσης λειτουργούν με αέρια και θα μπορούσαν να λειτουργούν με βιομάζα, αλλά δεν γίνεται προς στιγμή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ούτε μου αρέσουν όσα συμβαίνουν στις τρεις βαλτικές χώρες. Πέντε χρόνια, εκατομμύρια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τρεις βαλτικές χώρες δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για ένα κοινό, ε, ε, μια κοινή πλατφόρμα στη θάλασσα. Έχουν χαθεί τόσα εκατομμύρια. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένα ενιαίο εργοστάσιο μεταξύ των τριών βαλτικών χωρών. Ε, λυπούμε, ας μιλάμε, ε, λυπάμαι, ας, μιλάμε με γεγονότα όταν κάνουμε τέτοιε παρατηρήσεις. Και η δήλωσή σας η Ευρώπη να είναι πρώτη στις ανανεώσιμες. Σωστά θέλετε να διασυνδέσετε με την ενεργειακή ασφάλεια τις ανανεώσιμες. Όμως η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση τα τελευταία 10 χρόνια είναι η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία είχε 93% εξάρτηση από τι τις εισαγόμενες μορφές Τώρα έχει φτάσει το 80%. Γιατί, γιατί ανέπτυξε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει λοιπόν ένα στενό συσχετισμό μεταξύ των δύο, αλλά και άλλη μια διάσταση στις ανανεώσιμες. Η όλη διάσταση των εξαγωγών. Είμαστε ηγέτες στην αιωλική. Όμως ε, ο παγκόσμιος οργανισμός ενέργειας την έκθεση του την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε ότι η ολική και τα φωτοβολταϊκά είναι το μέλλον. Ε, και αυτό παρατήρησε. Εσεί, Επίτροπε, τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε η βιομηχανία των φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη που του ε, έχει αφήσει πίσω ε, το ντάμπινγκ των Κινέζων, οι οποίοι είναι και σε ανταγωνισμό με του Αμερικανού. 750 εκατομμύρια δάνειο για τα φωτοβολταϊκά δόθηκε την περασμένη εβδομάδα τη στιγμή που ερευνητικά κέντρα ε, στην Ευρώπη κάνουν παρόμοιες προτάσεις και ψάχνουν επενδύσεις και δεν, δεν τα πήρε η Ευρώπη τα, τα χρήματα αυτά. Δεν πρέπει λοιπόν τα φωτοβολταϊκά πάνελ να έχουν ένα μέλλον και στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να τα διασυνδέσουμε με το επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρώπης ώστε να μπορέσουμε να επανακάμψουμε στην αγορά. Διότι εάν δεν ε, έχουμε ούτε 20% φωτοβολταϊκά για την Ευρώπη, αλλά είμαστε πρώτοι στον εξοπλισμό και τα δίνουμε στους Αμερικάνους και τους Κινέζους, πού είναι η επιτυχία μας. Δεν είναι αυτό η σωστή προσέγγιση. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε συνάδελφε. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, αλλά σας παρακάλεσα να είστε σύντομοι. Γύρω στα δύο λεπτά όχι τέσσερα. Παρακαλώ λοιπόν, έχουμε ακόμα 11 συναδέλφους στο κατάλογο. Ο κύριος Κόφορτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να πω ότι για να, δοθ... να λυθεί το τριπλό αυτό δίλημα μεταξύ ενέργειας, οικονομίας και περιβάλλοντος είναι το πιο δύσκολο. Και για να το αποτύχουμε αυτό πρέπει να εστιαστούμε στην πράσινη οικονομία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ενεργειακά συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν εξετάζει πώς μπορούν να θερμαίνονται για παράδειγμα ολόκληρες περιοχές, πώς μπορεί να υπάρχει κοινό σύστημα ενέργειας επίσης ε, Ξέρουμε ότι η θέρμανση αποτελεί ένα μεγάλο τομέα κατανάλωσης της ενέργειας στην Ευρώπη και πολλά μπορούμε να κάνουμε για να μειωθεί το κόστος της ενέργειας και να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί και να χρησιμοποιούνται πιο πολλές ανανεώσιμες στο δημόσιο δίκτυο. Για το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Με τα εφιστάμενα δίκτυα ηλεκτροδότησης σήμερα, διάφορα κρατημέλη εμποδίζουν από την πρόσβαση στην αγορά και έτσι δεν υπάρχει ενιαία αγορά τι πρόκειται να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βράχει πρόθεσμα για την ε, οδηγία για το οικολογική σήμανση και την επισήμανση. Να πω ότι έτσι μπορούμε να σώσουμε και να εξοικονομήσουμε πολλή ενέργεια και είμαστε διτεθμένοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κατεύθυνση αυτή. Συζητήσατε επίσης το θέμα των κτηρίων. Σημαντικό και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Να ζητήσουμε από τα κρατημέλη να εκπληρώσουν τις υποχρέωσεις τους σε ό,τι αφορά και την οδηγία για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ευχαριστώ κύριε Βερικούνη, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε αυτή την ευκαιρία για αλλαγή απόψεων πριν αποφασίσετε για το πρόγραμμα εργασία σα στου κόλπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χρόνο. Θα ήθελα να σας ζητήσω το πλαίσιο του 2030 για την κλιματική πολιτική και για την ενεργειακή πολιτική και για τη ΓΕΑΙΛΟΚ. Ε, δεν είναι σαφέ στην παρούσα φάση κατά πόσο θα υπάρξει στόχο στι μεταφορέ για τι ανανεώσιμε, κατά πόσο θα συνεχιστεί αυτό και για μετά το 2020. Όλοι γνωρίζουμε ότι η θητεία αυτή ήταν ο βασικό ε, λόγο για τη συζήτηση ILOC. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση για την οδηγία ILOC στο Κοινοβούλιο και εκ παραλλήλου υπάρχει το νέο πλαίσιο χωρίς να υπάρχει σύνδεση με το πλαίσιο του 2030 και την νομοθεσία αυτή. Για τα επόμενα χρόνια. Υποσχεθήκαμε και αυτό αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξει καλύτερη ρύθμιση, καλύτερη νομοθεσία και παραλλήλου θέλουμε καλύτερη, πιο πολλές επενδύσεις στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να επενδύσουν λοιπόν οι επενδύσεις σε πράσινη ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις θα πρέπει να δούμε σε βάθος χρόνου και όχι μόνο τι θα γίνει σε δύο-τρία χρόνια. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, ε, μια παύση, ένα διάλειμμα σε ό,τι αφορά την οδηγία ILOC. Θα θέλαμε να ακούσουμε την απόψή σας. Ευχαριστώ, κύριος Herbert Ρόιλ, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, με ικανοποίηση άκουσα ότι είπατε ότι δεν θέλετε διαρκώ να κάνετε νέε προτάσει, αλλά καταρχά να κοιτάξετε πώ έχουν εφαρμοστεί ήδη οι φυστάμενε αποφάσει που έχουν ληφθεί. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω και το εξή, να δούμε και ποιε ήταν ο αντίκτυπο των αποφάσεων πέρα από το να έχουν εφαρμοστεί. Και Κατά δεύτερον, είπατε στην αρχή ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή ε, ε, επιχείρηση και τη ευρωπαϊκού οικονομικού κλάδου και ότι η βιομηχανία και οι τιμέ παίζουν βασικό ρόλο. Μετά όμως μιλήσατε επί μακρόν για τα πολιτικά μέτρα, για το κλίμα, για την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις ανανεώσιμες. Δεν πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε αν η μία ή η άλλη πολιτική απόφαση οδηγούν σε σπατάλες στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αν κάποια απόφαση οδηγεί σε υψηλές τιμές τη βιομηχανία και έτσι βλάπτει τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητά της και επίσης μήπως θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη καλύτερα κάποιες άλλες ενεργειακές πήγες στην Ευρώπη αντί να τις απαγορεύσουμε σε ό,τι αφορά το αέριο, τον άνθρακα. Πώς θα διαμορφωθεί λοιπόν το μέλλον και πώς μπορούν λοιπόν να προωθηθούν αποδοτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί μήπως το σύστημα που έχουμε τώρα είναι υπερβολικά δυσκίνητο και ακριβό και χρειάζονται ε, επιδοτήσεις διαρκώς. Κατά τρίτον, μιλήσατε για την οδηγία για την οικολογική σήμανση. Άκουσα ότι ο Γιούγκερ και το Επίτροπο Τίμερμαν ιδιαίτερο δήλωσαν ότι θα εξετάσουν τη ρύθμιση για να δουν κατά πόσο χρειάζεται τόσο πολύ ρύθμιση. Δεν πιστεύετε ότι σε θέματα οικολογικής σήμανσης χρειάζεται επίσης ένας τέτοιος έλεγχος, γιατί κατά πόσο είναι καν απαραίτητη η νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζωρίνιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση αυτή είναι στα πλαίσια του διαστρωμένου διαλόγου. Το πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε παρόλα αυτά είναι τομεακό. Καλό θα ήταν ε, ο αρχικός σας λόγος να περιληφθεί σε μια μπροσούρα και να μεταφραστεί σε 22 γλώσσες, διότι βάσει αυτού θα σας αξιολογήσουμε για το τι θα κάνατε την επόμενη χρονιά. Δεν θέλω να επαναλάβω όσα μόλις υπόθηκαν, απλώς να πω ότι στη Λίμα και μετά στο Παρίσι δεν θα συζητήσουμε μόνο για ένα ενεργειακό μοντέλο, ένα κοινό ενεργειακό μοντέλο που τίνει να αφανιστεί, ε, αλλά για ένα νέο κοινωνικό μοντέλο και ένα νέο οικονομικό μοντέλο ε, που θα πρέπει να συσχετιστεί με, τη με τον νέο πρότυπο για την κοινωνία. Εδώ ε, θα κρυθεί το μέλλον της Ευρώπης και ε, δεν θα θέλαμε να, να γίνει μια καρικατούρα αυτό το κοινωνικό μοντέλο που δεν μπορούμε πλέον εμείς να το επιβάλλουμε. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε άλλους. Ε, όταν μιλάμε για διασύνδεση, τι εννοούμε. Λέμε και ξαναλέμε διασύνδεση. Αλλά πού είναι ευφύ εδώ της Ευρώπη, πού είναι τα ευθύ δίκτυα, πού είναι η δυνατότητα τη βιομηχανία και τη κοινοτομία, γιατί δεν ε, καταφέρνουμε να ε, συνεισφέρουμε σε την αποδοτικότητα της αγοράς με όλα αυτά τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, τι μπαταρίε, του φορτιστέ, γιατί δεν έχει βρεθεί λύση. 80% της ενεργειακής αποδοτικότητας ακούσαμε ότι το πετύχαμε εμείς γιατί ακριβώς επενδύσαμε στην Πορτογαλία στις ανανόσιμες πηγές ενέργειας και επενδύσαμε στο εθνικό μας δίκτυο, ένα εθνικό δίκτυο με υποδομές πρέπει να αξιοποιήσουμε ό,τι βιομηχανική δυνατότητα ε, έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η καταπολέμηση λοιπόν της υπερθέρμανσης του πλανήτη πρέπει να οδηγήσει σε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Αυτά. Ευχαριστούμε κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε, αναφέρατε τη δημιουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς ε, όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Ξέρετε ότι προκύπτει μεταξύ των πολιτικών ομάδων στην Ήτρε μάλλον συμφωνία και θέλουμε να λειτουργήσει γρήγορα αυτή η πρόταση το αποθεματικό για να επηρεάσει και τη λειτουργία του ETS. Ελπίζουμε δηλαδή να είναι πολύ σύντομη η υλοποίηση ενό τέτοιου κανονισμού. Τώρα, για την δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, θα συμφωνήσω με τη συνάδελφο και τον Ντάρλινγκ. Είναι από τις αμεσότερες λύσεις... που χρειάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και το ζητεί και ο κλάδος... και οι κοινωνικοί εταίροι. Μιλήσαμε και για τη μείωση του κόστου της ενέργειας. Γι' αυτό ανησυχούν οι οικογένειε, οι τοπικέ κοινότητε, στη δική μου την επαρχία, τα βόρειο-δυτικά τη Αγγλία. Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα ζήτημα που πιέζει, πιέζει πολύ. Με ενδιαφέρει λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσετε, πώς θα ρυθμίσετε και θα βρείτε λύσεις για το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Ευχαριστούμε συνάδελφος Μαρτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας θέσω ερωτήσεις πολύ συγκεκριμένες και ακριβείς για να επιτύχετε τους στόχους που αναφέρατε προηγουμένως. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τα κριτήρια στοχοθεσίας. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της μόχλωσης και με τι προσέγγιση, με ευρωπαϊκή ή μήπω τελικά ποτέ έχουμε την ε, συγκέντρωση μιας, συστά, σειράς από εθνικά προγράμματα. Μιλήσατε για 15 75 ε, δις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Τι θα γίνει με την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων από τα 75 που, ε, δις που αναφέρατε θα αξιοποιηθούν ακριβώς για τα, έξοδα, τα τρέχοντα έξοδα της ε, βελτίωσης της θέρμανσης των κτηρίων. Βλέπουμε για το πρόγραμμα Juncker ότι έχουν γίνει πολλές ανακοινώσεις, αλλά τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν, να έχουν τελικά τα 21 που προβλέπονται για το αποθυματικό μπορεί τελικά να καταλήξουν αλλού. Ε, Ποιο θα είναι τελικά ο αντίκτυπο αυτού του προγράμματο σε πράγματα που ήδη έχουν ξεκινήσει από πέρσι. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι που είστε εδώ. Θέλω καταρχάς να σας ευχηστήσω την προσοχή ε, στο γεγονός ότι αυτή εδώ η Επιτροπή είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας. Και άρα όταν μιλούμε για βιομηχανία συχνά υιοθετούμε μία μανιχαϊστική στάση και αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι βιομηχανία από μόνη της. Βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν δεν υπήρχε βιομηχανία υψηλής εντάσεως ενέργειας, πάρα πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν, γιατί οι συνιστώσεις, τα συστατικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παράγονται από βιομηχανίες που χρειάζονται πολλή ενέργεια και είναι υψηλής εντάσεως ενέργειας. Αυτή λοιπόν η μανιχαϊστική, η μανιχαϊστική θεώρηση θα πρέπει να αποφευθεί, γιατί δεν μας οδηγεί πουθενά μας κάνει να έχουμε τεχνητά τείχη ε, στα οποία να προσκρούμε ξανά και ξανά. Επομένως, με αυτή την παραδοχή, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι βιομηχανίες που καταναλώνουν σε μεγάλη ένταση, ένταση ενέργεια θα πρέπει στην ανάπτυξή τους να έχουν ένα στοιχείο αποδοτικότητας και αυτό είναι ένα υπογραμμισμένο με όλους τους τόνους να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ενεργεία που καταναλώνουν. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό προσπαθεί να γίνει, αυτό προσπαθείτε να κάνετε στη στρατηγική άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν θα πρέπει να βάλετε μόνο τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Θα πρέπει κάποιο εδάφιο, κάποιο κεφάλαιο, κάποια διάταξη να ασχολείται μόνο με το κλάδο που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια μέσα σε όλη αυτή τη βιομηχανία. Θα πρέπει δηλαδή η ενεργειακή αποτελεσματικότητα να είναι προαπαιτούμενο, να είναι θέλετε, κριτήριο και για τη βιομηχανία. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει τέτοιο στοιχείο στο κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρο μα τώρα. Μία ερώτηση μόνο έχω να σας κάνω, κύριε Επίτροπε. Ο κύριο Έγκελ. Πιστεύετε πραγματικά ότι η κοινή ενεργειακή αγορά είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι δυνατό αν κάθε χώρα αποφασίζει για το ενεργειακό της μείγμα. Σας ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε, τι γίνεται με την ΕΚΟΓΑΣ. Δεν είναι πια ισπανική επιχείρηση. Ήταν μια επιχείρηση πολύ καινοτόμα για τις, ε, τους σταθμούς ε, θερμικής επεξεργασίας που οδηγούν σε καθαρό άνθρακα και εντάσσονται σε όλη αυτή τη ε, διαδικασία της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Είναι μια πολύ καινοτόμος επιχείρηση, πρωτοπόρος και στην Κίνα και στη ΣΥΠΑ και αλλού. Είχε 50% κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 50% από εθνικά κονδύλια. Είναι βιώσιμη επιχείρηση, το λένε και οι ίδιοι τις ο ισολογισμός του 11 και του 12 ήταν θετικός, τα αποτελέσματα ήταν θετικά και πηγαίνει προσκλήσιμο κλείσιμο δυστυχώς ευθύς αμέσως. Κυρίως για τρεις βασικές αιτίες. Πρώτον, αλλάζει η κατανομή της ενέργειας, δεν μπαίνει στο ειδικό καθεστώς, μπαίνει πλέον στο συμβατικό καθεστώς. Ζητείται το Δεκέμβριο το σχετικό βασιλικό διάταγμα και η έγκριση και ψήφισή του για ότι υποτίθεται ότι πρέπει να χρησιμοποιεί άνθρακα που έχει ε, παραχθεί στη χώρα και για διάφορους άλλους τέτοιους λόγους. Λοιπόν, υποτίθεται ότι πρέπει να προωθήσουμε τέτοιου είδους τεχνολογίες και να τις ρυθμίσουμε. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις που είναι βιώσιμες με υψηλή προστιθεμένη αξία. Είναι κρίμα να κλείσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο Γκομπάτσικ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Να πω κάποια πράγματα για τις τιμές της ενέργειας. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. πιστεύω στην ε, λογική, την ορθολογιστική σας προσέγγιση ότι πρέπει να συνδυάσουμε την νομοθεσία. Όμως αυτά που μας λέτε δεν φαίνονται και πάρα πολύ διορατικά. Μιλήσατε για τους διασυνδετές και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε αρκετά κονδύλια για να τους φτιάξουμε για σκοπούς διασύνδεσης. Ή μετά ε, μιλήσατε για κάποιες πηγές ενέργειας, συγκεκριμένα χώρες όπως η μετα Είναι ένας αναξιόπιστος ε, προμηθευτής η Ρωσία. Βλέπουμε τι σοβαρές δυσκολίες και τελικά σε απαιτεί αποτυχία κατέληξε το εγχείρημα του Ναμπούκο. Οπότε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως ήρθε η ώρα να ξαναδείτε τον άνθρακα. Ακούσαμε για το CCS, δηλαδή την δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, ακούσαμε για νέους τρόπους ε, που μπορεί να καίγεται ο άνθρακας χωρίς να προκαλεί τους ίδιους ρήπους, ακούσαμε για το σχιστηλιθικό αέριο και το υγροποιημένο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε μας έδειξαν ότι μπορεί να παράξει κανείς ε, υγροποιημένο σχιστολιθικό αέριο σεβόμενο το περιβάλλον. Δεν πρέπει αυτά τα θέματα να τα ξαναδούμε και να αναπτύξουμε βιομηχανικέ λύσει βάσει τέτοιων πηγών ενέργεια που επιτρέπουν φτηνότερε τιμέ. Ευχαριστούμε κύριο Σιλικιώτη. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, εγώ θα επανέλθω ε, στο θέμα του νότιου διαδρόμου για ενίσχυση τη ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη. Ο νότιο αγωγό ματιώθηκε. Η νοτιοανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζει επίγουσε ανάγκε λόγω και τη κρίση στην Ουκρανία. Προβλήματα ενεργειακή επάρκεια ε, διαπιστώνονται και ευρύτερα, θα έλεγα, σε ολόκληρη την Νότια Ευρώπη. Είναι στι προτεραιότητε σα η ανάπτυξη ενό μεσογειακού κόμβου μέσω διαδρόμου από την νοτιοανατολική Μεσόγειο προ την Ευρώπη. Ε, τέθηκε και με ένα διαφορετικό τρόπο προηγουμένω το ερώτημα, χωρί να απαντήσετε συγκεκριμένα. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα πράγμα συγκεκριμένο όμω. Τι τελευταίε μέρε έρχεται στην ατζέντα μια κοινή πρόταση από τι ε, από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα για τη δημιουργία ενός αγωγού που θα ξεκινά από το Ισραήλ και την Κύπρο και μέσω Ελλάδα να έρχεται στην Ευρώπη ε, για να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικές ανακαλύψεις κοιτασμάτων τα τελευταία χρόνια ε, και στην Κύπρο αλλά και στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πώς αντιμετωπίζετε ως Επιτροπή ε, αυτό το θέμα ε, και αν υπάρχουν κάποιες σκέψεις ε, για τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου που θα ε, στηρίξει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ιδιαίτερα την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Νότια Ευρώπη ευρύτερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. 30 seconds for you, Tom. Σας ευχαριστώ. 30 δευτερόλεπτα έχετε, στον Μπουράνο. αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ σύντομα. Ναι, θα είμαι συνοπτικότατος. Επίτροπε, μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη συνεννόηση, διότι στην ε, Ιταλία ένας, μιλήσαμε για φόρο για τον άνθρακα βάσει της παραγωγής ε, εκπομπών και την θερμοδυναμική ε, περιεκτικότητα. Όχι για οικολογικό φόρο όμως. Αυτό θα ήταν περίεργο να το προτείνουμε εμείς. Ευχαριστούμε. Επίτροπε, τώρα έχετε μια σειρά από παρατηρήσεις και ερωτήσεις πάλι. Θα σας παρακαλέσω να απαντήσετε σύντομα τις ερωτήσεις. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι οι κανόνες για τη διακυβέρνηση θα παρουσιαστούν στο πρώτο εξάμεινο του 2015, αυτό έχουμε αποφασίσει, και άρα οι όροι της διακυβέρνησης είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθήσουμε τον βαθμό στον οποίο κάθε κράτος μέλος τηρεί τις δεσμεύσεις του, έτσι ώστε οι συνολικές δεσμεύσεις να υλοποιηθούν. Να σας πω επίσης ότι Πρέπει να κάνουμε μελέτες αξιολόγησης αντικτύπου για το σύστημα εκπομπής ρήπων αναπεδιο, ανακλάδο, ανά ο οποίος ο καθένας έχει την περιπλοκότητά του και πρέπει οι αξιολογήσεις να γίνουν σωστά για τον εκάστοτε κλάδο και να δούμε ποιες είναι οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των αποφάσεων που λαμβάνουμε επιβάλλοντας τους κλάδους την χ και την ψη υποχρέωση. Τώρα, ως προς τον κύριο Ρόιλ. Είπατε ότι πρέπει να προβληματιστούμε για το κατά πόσο ορισμένες πολιτικές αποφάσεις είναι αυτές που ρυθμίζουν τις τιμές. Απαντώ λέγοντας ότι πάρα πολλοί είναι οι παράγοντες που εμπλέκονται στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας και πρέπει να τους δούμε όλους αυτούς τους παράγοντες, όλους. Ε, μερικές φορές οι κλάδοι είναι αδύνατο να ε, συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους. Μερικές φορές υπάρχει ανάδοχος μοναδικού προμηθευτή. Μερικές φορές υπάρχει έλλειψη διασύνδεσης. Ε, είναι πάρα πολλοί και πρέπει όλα αυτά τα εμπόδια να καταρριφθούν. Υπάρχει και το co-design. Πολύ συχνά έχουμε οδηγηθεί σε πολύ σημαντική οικονομική εξοικονόμηση. Δεν μιλάω μόνο για το πολύ αφιερεμένο ή πολύ ίσονο σημασία, αν θέλετε, παράδειγμα του προϊόντος του τηλέφωνου, του ντους, το με το οποίο ρυθμίζουμε τη ροή του νερού που βγαίνει και έτσι έχουμε εξοικονόμηση. Μιλάω για πολύ σημαντικά, ε, σημαντικούς τρόπους εξοικονόμησης. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος προτού εγκριθεί το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτές είναι οι γενικές γραμμές δράσης και ε, με αυτόν τον τρόπο θα προσεγγίσουμε την κατάσταση. Ως προς τη διάσκεψη ε, της Λίμας και των Παρισίων, αυτό το οποίο θα αναζητήσουμε είναι δέσμευση υποχρεωτική για τη μείωση των εκπομπών σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε η θερμοκρασία να μειωθεί. θα κάνουμε ε, θα υιοθετήσουμε δέσμευση για να μην υπάρξει θέρμανση, υπερθέρμανση άνω των δύο βαθμών Κελσίου, κάτι το οποίο θα ε, δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Ε, μίλησε ο βουλευτής κύριος Κρίφιν για το κατά πόσο μπορούν να τεθούν σε ισχύ το 2017 και όχι αργότερα όλοι αυτοί οι μηχανισμοί. Νομίζω ότι όσο πιο γρήγορα στείλουμε τα κατάλληλα μηνύματα στη βιομηχανία και σε όσους επινοούν και δημιουργούν καινοτομία, τόσο το καλύτερο. Το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι τα έργα που έχουμε δρομολογήσει δεν έχουν φτάσει σε επαρκές επίπεδο ορίμανσης. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να προωθούμε έργα που θα αποδεικνύουν σε μεγάλη κλίμακα ότι είναι εφικτό να μειωθεί το κόστος και ότι υπάρχει επαρκής ε, προμήθευση. Πρέπει να επενδύσουμε στις ε, υποδομές διασυνοριακών μεταφορών, να έχουμε καλύτερη και περισσότερη γνώση της πραγματικής χωρητικότητας του πόσο τελικά μπορούμε να αποθηκεύσουμε διοξίδιο του άνθρακα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε το γεωγραφικό του εντοπισμό. Πού είναι οι πηγές και πού είναι οι χώροι δέσμευσης και αποθήκευσης. Ο άνθρακας θα είναι σημαντικός και πρέπει να βρούμε τεχνολογία που να μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε άνθρακα στις μέγιστες και καλύτερες δυνατές ενεργειακές συνθήκες και να έχουμε και το σύστημα εκπομπής ρήπων, να έχουμε σωστή δέσμευση αποθήκευσης. Στις συμφωνίες που έχουμε με την ΕΠΑ και την Κίνα χρηματοδοτούμε μεγάλα έργα για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα για να δούμε κατά πόσο τεχνικό είναι βιώσιμα και οικονομικό είναι βιώσιμα. Και ε, θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τι άλλο έχω κύριε Πρόεδρε, κυρία Καστίγιο είπε ότι δεν πρέπει να ε, ξεχάσουμε ότι εδώ είναι Κοινοβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανίας. Συμφωνώ, αλλά τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη βιομηχανία και δεν είναι μόνο κίνδυνος, είναι και ευκαιρία. Είναι μεγάλη ευκαιρία οικονομική ανάπτυξη για τη βιομηχανία, η π.χ. ενεργειακή αποδοτικότητα και πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι, ηγέτε στον τομέα και στα φωτοβολταϊκά και στην νεολική ενέργεια. Στο σχέδιο Juncker ένα σημαντικό κεφάλαιο είναι η καινοτομία Πολύ έχετε αναφερθεί στο σχέδιο Γιούγκερ. Να σας πω λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης υποδομών διασύνδεσης και ε, επικοινωνίας μεταξύ των ΜΕΝ και των ΔΕ. Έχουμε δυνατότητες για μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα σε κτίρια, σε βιομηχανίες, σε διάφορα, πολλά και διάφορα πεδία. Και έχουμε και δυνατότητα να έχουμε καινοτομία, ανάπτυξη, σε αυτά τα πεδία. Θα έχουμε πολλαπλασιαστές με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα κράτη-μέλη θα υποβάλουν ένα σακούλι έργων, αν θέλετε, και θα εξαρτηθεί από το κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει το ίδιο ποιο ε, κλάδο θέλει να αναπτύξει. Άλλα κράτη-μέλη θα στοιχηματίσουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα, άλλα θα πρημοδοτήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άλλα τις ευρυζωνικές συνδέσεις εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας ε, κτλ το ενεργειακό μείγμα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και αυτό λέγεται ξεκάθαρα. Δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δρομολογήσει τα πάντα έτσι ώστε ό,τι και αν επιλέξει το κράτος μέλος να μπορέσει να το αναπτύξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να έχει ε, όσο το περισσότερες εγγυήσεις περιβαλλοντικής ασφάλειας ή επάρκειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ενεργειακό μείγμα είναι απόφαση του κράτους μέλους. Για να αλλάξει αυτό πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες. Έγινε λόγος από τη Συρία Ακαβεθών για τις επιχειρήσεις και για την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν είναι εύκολο να νομοθετήσουμε. Θα το διερευνήσουμε κατά πόσο είναι δυνατόν να νομοθετήσουμε και να προτείνουμε νομοθεσία για αυτό το θέμα. Καθοριστικός παράγοντας είναι το σύστημα κατανομής, το διανεμητικό σύστημα και αυτό είναι κρατική αρμοδιότητα. Φιλοδοξούμε στην αγορά τα συστήματα κατανομής χωρητικότητας και δυναμικότητας να ε, εξισωθούν, αν θέλετε να εξομοιωθούν. Αυτό θα το καταφέρουμε όσο περισσότερο πάμε σε μια ενιαία εσωτερική αγορά ενέργειας. Ίσως δεν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη σε αυτές που, για όσους δεν κατάφερα να απαντήσω στην ερώτησή τους. Βλέπετε τι χαμός γίνεται εδώ με τα χαρτιά, πόσο λίγο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Πιστεύω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Όπως είδατε είχαμε τις, την ακρόασή μας, είχαμε την τακτική μας συνεδρίαση, πλήθος ερωτήσεων. Ήταν η πρώτη μας ε, ε, επαφή με την Επιτροπή από τη στιγμή που ανέλαβε την θητεία του. Σας ευχαριστούμε πολύ Επίτροπε λοιπόν για την προθυμία σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε ένα λεπτό θα ξεκινήσει η Χριστουγεννιάτικη δεξίωση, αλλά να πω το εξή. 9 το πρωί. 9 το πρωί δεν χρειάζεται να είστε εδώ. Μόνον οι συντονιστές. Καλές ειδήσει. Μόνον οι συντονιστές τη 9. Στις 10 οι υπόλοιποι. Μην ξεχάσετε τις κάρτες σας, ψηφοφορίες στις 10 ψηφοφορίες και τα επόμενα σημεία. Τα λέμε αύριο το πρωί. Είσαι ένα λεπτό. Ευχαριστώ, γεια σας.